Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, δεν έχει ζητήσει κανείς κάποια αλλαγή, οπότε υποθέτω πως εγκρίνεται μετά να σας πενθυμίσω πως ο συνήθως η συνεδρίαση μας μεταδίδεται ζωντανά και περνάμε στο επόμενο θημείο απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης του 9 ου και 10ου εισηγητής ο Μάρτιν Έρενχάουζερ και έχουμε ανταλλαγή απόψε με εκπρόσωπο των Τάμζιν Μπάρτον, δηλαδή Γενικό Διευθυντή για τις δραστηριότητε εκτός της Ένωσης, ε, τον οποίο καλώς ορίζω και αν συμφωνεί και ο εισηγητής θα ήθελα πρώτα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, Ήθελετε να πείτε κάτι εσείς, όχι. Όχι. Τότε κατευθείαν τον λόγο έχει ο κύριος Μπάρτον. Καλώς ήρθατε και έχετε τον λόγο και καλημέρα κιόλας. Thank you very much uh, for the warm welcome. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό καλωσόρισμα. Ήρθα πριν από ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο και τότε ήμουν νέα στη θέση μου. Ελπίζω να έχω μάθει πολλά έκτοτε και να μπορώ να είμαι σε θέση να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ίσως ε, θεωρήσετε ότι δεν είμαι σε θέση να, τα πω όλα για τα πάντα, αλλά θα έλεγα εν είδη εισαγωγή ότι έλαβα σοβαρά υπόψη ε, κάποια από τα σχόλια που κάνατε την περασμένη φορά και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας δείξω ότι σημειώθηκε πρόοδος από πέρσι. Επίσης, έχετε συμβάλει κι εσείς ε, ώστε η δανειοδοτική δραστηριότητα σε σχέση με τις χώρους, τις γειτονικές χώρες εταίρους μας ε, να ευοδοθεί. Πέρσι είχαμε ακούσει και τους ε, ειδήμονες από το οικονομικό τμήμα και τις σχετικές υπηρεσίες και τους ζητήσαμε να συστήσουν ένα νέο πλαίσιο δραστηριοτήτων όπερ και έγινε και ελπίζω να πάρετε τώρα ένα φυλάδιο που έχουμε προετοιμάσει για να σχηματίσετε κι εσείς μια εικόνα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί βάσει του νέου πλαισίου. Ε, προσπαθήσαμε να εκπονήσουμε τη νέα μέθοδο και να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε τους ανθρωπίνους και άλλους πόρους μας, κυρίως επειδή πρέπει να δρούμε σε συνέργεια με άλλους. Ε, εμπλακήκαμε λοιπόν ε, σε ομάδες εργασίες ε, με εκπροσώπους άλλων διεθνών οργάνων. Φυσικά διαβουλευτήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθώντας να εκπονήσουμε κάτι ευεφάρμοστο, απλό και που δεν συνεπάγεται μεγάλο άχθος για τους δανειστές, αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε δηλαδή, καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες. Χρησιμοποιείται το νέο πλαίσιο, αλλά φυσικά θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν τα προγράμματα που θα τρέξουν βάσει του νέου πλαισίου. Θα δείτε λοιπόν εν καιρό τα αποτελέσματα, όχι ακόμα. Στο ενδιάμεσο διάστημα και δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχετε για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, ε, συζήτησα με τους συναδέλφους από το τμήμα επικοινωνίας ε, και το τμήμα επιχειρήσεων και προετοιμάσαμε άλλο ένα φυλάδιο για να ε, ε, σχηματίσετε μια σφαιρικότερη εικόνα σε σχέση με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε αυτά τα δύο φυλάδια κανονικά στη διάθεσή σας και ελπίζω ότι θα συνειδητοποιήσετε ε, ότι αυτή την επιχείρηση την αναλάβαμε κατόπιν του δικού σας αιτήματο ε, εν πωλής, οπότε χαίρομαι που μπορώ να σας το ανακοινώσω σήμερα. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τομείς που σχολιάσατε πέρσι, αν θυμάμαι καλά, και θα μπορούσα να σας ε, περιγράψω την διάμεση τάξη πραγμάτων, την πρόοδο που είχε σημειωθεί. Ο κ. Σίμψον, παραδείγματο χάρη, είχε ρωτήσει πολλά για την πολιτική καταπολέμηση της απάτης είναι ένας τομέας ε, όπου όντως σημειώθηκε πρόοδος ε, και θα το σχολιάσω. Επίσης αναπτύξαμε ένα νέο πιλωτικό σύστημα που θα μας βοηθήσει να συνεργαζόμαστε καλύτερα με άλλους συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να έχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντονεί εγκλήματα ε, και με τα αρχεία η εμπειρία δείχνουν, δείχνει ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Επίσης ε, θα μπορώ να σας πω κάποια νέα για τον αξιωματούχο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα αρμοδιότητα μα ε, που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Το EDPS φυσικά έχει σχέση με αυτό και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό μπορεί να βλάψει κάποιες επιχειρήσεις όταν υπάρχει μόνο υπόνοια, υποψία και όχι ε, κάτι αποδεδειγμένο. This month we should have uh, a view from the EDPS. Uh, this time next year about how that's actually working or if any of you θα ε, έχουμε και επίσκεψη του υπόπτη προσωπικών δεδομένων. Ε, πέρσι στο Λουξεμβούργο υπήρξε μια άτιμη, άτυπη επίσκεψη και θα έχετε τη δυνατότητα σε μελλοντική συνεδρία να θέσετε και άλλες ερωτήσεις σε σχέση με τις δραστηριότητε του υπόπτη. Ε, σε σχέση τώρα με το μηχανισμό διευκόλυνση των επενδύσεων, ε, κάναμε κάποιε προσπάθειε ε, να επαναπροσανατολίσουμε το σύστημα για να καλύψουμε τι ανησυχίε σα. Όπω ξέρετε, βεβαίω, έχουμε καθυστερήσει ένα χρόνο, διότι βλέπουμε την έκθεση για το 2010 και όχι για το 2011 και πιστεύω ότι μόλις λάβουμε και την έκθεση για το 2011 θα διαπιστώσετε ότι έχουν σημειωθεί και άλλες αλλαγές. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Ε, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις ε, ε, έχετε. Έχουμε στη διάθεσή μας και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που μπορούν να συμπληρώσουν αν δεν μπορούν να απαντήσω σε όλα. Έχουμε και ένα συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπάρξουν ερωτήσει σε σχέση με τη συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο πάντως ε, ε, ε, σημειώθηκαν πολύ θετικέ εξελίξει στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουμε την εξωτερική εντολή και την αναδιαπραγμάτευση τη Συμφωνία Κοτονού ε, και ε, ε, με τη βοήθεια και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η συνεργασία μας και αυτό είναι και ένα από τα βασικότερα επιτέγματα από το που ανέλαβα εγώ τη θέση. Σας ευχαριστούμε κυρία Μάρτιν. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη συνεργασία μας μέχρι στιγμής. Ζητήματα που έθεσα πάντα τα απαντούσε αμέσως και ικανοποιητικά ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά έχω έτσι μερικές ερωτησούλες για σας σήμερα. Να ξεκινήσω με τις ροές, τις χρηματικές. Από ό,τι κατάλαβα τα κράτη-μέλη πληρώνουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης πληρώνουν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που πληρώνουν μετά τις κοινοπραξίε. Οι κοινοπραξίε πληρώνουν τους εταίρου και οι εταίροι πληρώνουν τα έργα. Πολλές τράπεζες υπάρχουν ενδιάμεσα. Και χρεώσεις και το και Και πρώτα γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαδρομή του χρήματος. Δεύτερον, υπάρχουν προτάσεις για να μειωθεί κάπως αυτή η αλυσίδα. Τρίτον, με τις τράπεζες αυτές τις ενδιάμεσες έχετε κάνει καν, καμιά συμφωνία για τα επιτόκια και για τις ε, κοινοπραξίες αυτές και τους τέρους ε, που πρέπει και αυτοί βεβαίως να λαμβάνουν τα λεφτά ε, αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις ε, διοικητικές ε, δαπάνες. Επίσης, όπως είπα, υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες που αναμειγνύονται και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο κριτήριο ιδιοκτησίας των τραπεζών ανευρωπαϊκές αμερικάνικες γιατί πρέπει βεβαίως να ενισχύονται και οι ε, τράπεζες οι τοπικές. Μετά η υπόθεση πόρη. Η ΜΚΟ Counterbalance ανέφερε την υπόθεση ότι πληρώνονταν σε νιγηριανές εταιρείε λεφτά παρά το ότι οι διοκτήτες τους ήταν ύποπτοι διαφθοράς. Και ο κύριος Ολόπκο μετά που είναι κατά της διαφθοράς απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, με, ζητώντας ε, να συναντηθεί ε, μαζί τους και όχι μόνο αρνήθηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά έδωσε και την ταυτότητά του στις Νιγηριανές αρχές. Τα ερωτήματα μου είναι πρώτον ισχύει αυτό και δεύτερον πράγματι γνωστοποιήσατε την ταυτότητά του στις αρχές της Νιγηρίας. Αυτά από αυτή την πλευρά για το επόμενο ερώτημα για τους τελικούς δικαιούχους και εκεί πέρα δεν ξέρω αν έχετε έλεγχο ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι και που καταλήγουν τα λεφτά. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν για να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους και τη δεύτερη επιμέλεια πρέπει να δείχνετε και την παρακολούθηση αυτών των πραγμάτων. Και τελευταίο ερώτημα όσον αφορά την μονάδα καταπολέμησης της απάτης η οποία έλαβε 45 καταγγελίες το 2009 και 82 καταγγελίες το επόμενο έτος. Μιλάμε σχεδόν για διπλασιασμό. Πού οφείλεται αυτό και δεύτερον σε ποιο βαθμό τα ε, κονδύλια του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Ανάπτυξης επηρεάστηκαν από αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Ρενχάουζερ. Να ρωτήσω τώρα τις ομάδες. Ε, έχουν να πούν τίποτα στον πρώτο αυτό γύρο. Όχι. Να δώσω λοιπόν στην κυρία Μπάρτον. Α, με συγχωρείτε. Ε, Μιούλερ και μετά κυρία Ιβάνοβα. Έχω ένα ερώτημα που δεν έχει καμία σχέση με την ε, γενική εισήγηση και απολογισμό, όλα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όπου η μία χώρα μετά από την άλλη υποβαθμίζεται από τη Standard Poor's, από τη Moody's και όλους τους άλλους οίκους αξιολόγησης. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει εγγύηση όπως προς την κεφαλαϊκή επάρκεια της ΕΤΕ και των άλλων τραπεζών. Δηλαδή, τι προβλέπετε για την ΕΤΕ. Και μιλάμε για κεφάλαια τα οποία ε, την χάνουν εγγύησης από τον προϋπολογισμό. Εάν υποβαθμιστεί η ΕΤΕ, ίσως υπάρχει ε, επιρροή στις δυνατότητες δανειοδότησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το σύστημα εποπτείας και ελέγχου έχουμε την ανάλυση του ελεκτικού συνεδρίου που αναφέρει ότι για τέταρτο συνεχόμενο έτος το σύστημα εποπτείας και ελέγχου είναι, ε, καλύπτει τις ανάγκες μερικώς, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Ως προς τους δικαιούχους, έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα να σας δώσω αλλά θα το υποβάλω στο επόμενο τμήμα των συζητήσεων. Ευχαριστώ. η Ja, ähm, Ευχαριστώ. Μετά από αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω πως εγώ διάβασα ότι προσφάτως το σύστημα των μικροδανείων, τουλάχιστον έτσι διαβάσαμε στη Γερμανία. Και τώρα... Δεν θέλω να πω να χαρακτηρίσω τα πράγματα, αλλά οι μεγάλες προσδοκίες που είχαμε, ειδικά στην Αφρική και στην Ασία, ε, δεν ε, δόθηκαν. Είπα, μάλλον υπάρχουν αμφιβολίες για τη σχέση κόστους-οφέλους, ειδικά στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν το συζητάτε κι εσείς και αν το συζητάτε όπως συζητείτε αυτή τη στιγμή στο γερμανικό τύπο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βάιλερ, δεν βλέπω κανέναν να ζητάει το λόγο, οπότε μπορώ κι εγώ. Ναι, βεβαίω. Ο κύριο Λιμπεράτσκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο ε, διότι δεν θέλω να συζητήσουμε εδώ για οικονομικές δραστηριότητε. Πέρα από τα οικονομικά και τα κοινωνικά θέματα, θα ήθελα να ακούσω αν έχετε κάποια άποψη περί της διαφάνειας της προβολής ε, του έργου σας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνεται η εντύπωση ότι κάνουμε κάτι καλό, δημιουργούνται θετικά συναισθήματα στους πολίτες και στις χώρες όπου βρίσκονται οι δικαιούχοι για την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ίδια την Ένωση. Σας ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ακούσουμε την απάντηση της ΕΤΕ. Κυρία Μπάρτον. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ε, για κάποιες ερωτήσεις ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων διότι δεν τις έχω κατανοήσει πλήρως. Ε, θα συνδέσω το τελευταίο με το πρώτο ερώτημα. Με ρωτήσατε για τις ε, ροές ε, χρημάτων ε, του Ταμείου σε διάφορα επίπεδα. Ουσιαστικά μιλάτε για τους εταίρους της Ένωσης για τη χρηματοδότηση. Από ό,τι καταλαβαίνω πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπούσε ακριβώς την προβολή του έργου μας και δικαίως το θέτετε κι εσείς κατά πόσο προβάλλεται το έργο δηλαδή εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής ε, θεωρώ εν γέννη ότι η ΕΤΕ ακόμη και μέσα στην Ένωση δεν είναι επαρκώς προβεβλημένη, ίσως ε, γιατί είχαμε εστιάσει στο να έχουμε απτά αποτελέσματα από το έργο μας ε, και να διαχειριζόμαστε σωστά τους πόρους μας, καλύτερα να διαχειριζόμαστε τους οικονομικούς πόρους δηλαδή από ό,τι την εικόνα μας μπορούμε να αυξήσουμε την επικοινωνιακή προβολή των δραστηριοτήτων μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμφίβολα ε, και μπορούμε να ε, βασιστούμε σε αυτά που ήδη έχουμε καταφέρει και σας παραπέμπω και πάλι σε αυτό το φυλάδιο όπου έχετε πληροφορίες ε, και πριν από λίγο το Σεπτέμβριο θυμάμαι καλά ε, μαζί με τον Επίτροπο Πίμπαλξ επισκεφθήκαμε την Νότιο Αφρική, έγινε μια μικρή τελετή για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα ε, που ολοκληρώθηκε στην Νότια Αφρική. Ε, πρόκειται για μια επιχείρηση startup. Ε, όλα τα προγράμματα εκεί πέρα τους ή άλλως είναι επιχειρηματικού κινδύνου και σχετίζεται με όσους βρίσκονται σε δυσμενή θέση μετά και το καθεστώς του Απαρτχάιντε και Ε, πιστεύω ότι κάναμε τη διαφορά, όχι μόνο μας φυσικά, γιατί συνεργαστήκαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βοηθήσαμε ούτως ώστε να χορηγούνται καλύτερες υπηρεσίες υγειονομικής ε, και ατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτά για το τελευταίο, αλλά για το πρώτο ερώτημά σας, για τους ε, μεσάζοντες, τους διαμεσολαβητές, όλη αυτή την αλυσίδα. Ε, κοιτάξτε, είναι, πρόκειται για μια μεγάλη οργάνωση και οι εκεί ο οργανισμοί δεν έχουν τόσο ευρία δραστηριότητα, αλλά πιστεύω ότι ε, όλοι μπορούν να ε, συμβάλλουν ε, ώστε να στηρίξουν διάφορα τέτοια προγράμματα που πάντοτε υλοποιούνται σε συνεργασία διαφόρων εταίρων, όπως σας έλεγα. Ε, έχουμε διαδικασία αξιολόγησης από τους ομότιμους, συντονίζουμε τη δράση διαφόρων εταίρων μας ε, και όντως αυτό συνεπάγεται ένα επιπλέον στρώμα ε, που δεν μας επιτρέπει με ευκρίνεια να δούμε ακριβώς με ποιο τρόπο διοχετεύονται ε, και πού τα κονδύλια της ε, ΑΤΕ, αλλά πρέπει να συντονιστούν, ε, ξέρετε, οι δράσεις τόσων πολλών οργανισμών. Τώρα, σε σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία και πάλι, είναι προφανές ότι θα θέλαμε όλοι κατευθείαν να δίνουμε σε αναπτυσσόμενες χώρες τα λεφτά στους ενδεείς και να δούμε τι, ποιο αποτέλεσμα θα έχουν, αλλά ξέρετε ότι στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό και είναι δύσκολο τόπου να έχουμε εποπτικό και ελεγκτικό μηχανισμό ε, αν ακολουθούσαμε ένα τέτοιο σύστημα. Άρα χρειαζόμαστε πιο περίπλοκες δομές ε, με σαφείς κανόνες και κατάλληλη εποπτεία και αυτό ακριβώς και έχουμε, εφαρμόζουμε πάντοτε σαφέστατα κριτήρια επί τη βάση των οποίων επιλέγουμε τις ε, τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για εταιρική διακυβέρνηση, για κοινωνική ευθύνη. Υπάρχουν ε, αυστηρά κριτήρια ως προς την προληπτική εποπτεία επίσης ε, και για όλα τα προγράμματα φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας αν θέλετε όπως αν πρόκειτο για ένα παγκόσμιο δάνειο σωστό έλεγχο, σωστή εποπτεία. Επίση, ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ε, προστιθέμενη αξία, δηλαδή να βρούμε την ισορροπία. Όντω, ο δικαιούχο να υποφελείται από το δάνειο, αλλά ε, χωρίς ε, να δίνουμε υπερβολικά χρήματα εκεί όπου δεν χρειάζονται, ανακόπτοντας έτσι την ανάπτυξη, γιατί υπάρχει υπερκορεσμός ε, της αγοράς. Και άρα πρέπει να γίνεται και σύνδεση με την εποπτεία και τον έλεγχο για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και να επιτυγχάνουμε αυτή την λεπτή ισορροπία, ούτω ώστε να είναι απτά και τα ωφέλη για τους δικαιούχους, αλλά και γενικότερα. Αυτά θα έλεγα σε σχέση με το πρώτο ερώτημά σας και πιστεύω ότι μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να το συζητάμε και όλη μέρα. Uh, uh, Για την εταιρεία Counterbalance και τις κατηγορίες ε, στην περίπτωση αυτή απάτη στην Ιγυρία, ξέρετε δεν γνωρίζω προσωπικά αυτή την υπόθεση, γνωρίζω πολύ καλά ε, την οργάνωση Counterbalance ε, γιατί τακτικά έχουμε διάλογο μαζί τους χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε όλοι, και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Ε, εξετάζει, παρακολουθεί, αν θέλετε, τις δραστηριότητες ε, της ΕΤΕ. Πολύ καλό είναι να έχουμε με κυβερνητικές οργανώσεις που ελέγχουν τις δραστηριότητες ε, και μας, με τη δράση τους και το άγρυπνο βλέμμα τους μας επιτρέπουν να έχουμε υψηλά κριτήρια, αλλά περιορίζεται η αποτελεσματικότητα της counterbalance όταν εστιάζεται μόνο στην ΕΤΕ και δεν βλέπει την σφαιρική σφαιρικότερη εικόνα, παραδείγματο χάρη, αν συγχρηματοδοτήσουμε με άλλου οργανισμού. Η counterbalance δεν λέει τίποτα για του υπολείπου ε, και ε, διαπιστώσαμε ότι οι ισχυρισμοί τους ε, δεν ευσταθούν όταν ακολουθεί έρευνα συχνά. Ε, μας δίνουν εκθέσεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει πλήθος ανακριβών στοιχείων ε, μέσα. Τέλος πάντων έχει προχωρήσει ο διάλογος με αυτήν την οργάνωση και τελευταία έκθεση που νομίζω δημοσιεύτηκε χθες ε, αναφέρει, α και είχαν και την ε, ευγένεια να μας τη δώσουν και νωρίτερα την έκθεση για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να ε, τους ε, στήσουμε την προσοχή σε αυτά τα ανακριβή στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχουν διορθωθεί, αλλά τουλάχιστον μας έδωσαν την ευκαιρία να το κάνουμε. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη κατηγορία ε, δεν δύναμε να σας δώσω μια απάντηση, αλλά μπορώ γραπτός να σας την στείλω, πάντως γενικά. Ε, υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί που ε, δεν προκύπτουν από ε, ξενυχιστικού ελέγχους. Υπήρχαν κάποιοι ισχυρισμοί σε σχέση με υποστηρίξη προγραμμάτων στην Αίγυπτο, παραδείγματο χάρη Ε, και ε, υπήρχαν κατηγορίες, μετά διαπιστώθηκε αυτά τα προγράμματα έτρεχαν υπό το προηγούμενο καθεστώς. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις για αυτή την υπόθεση την οποία γνωρίζω. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε διάλογο με ένα ευρύ φάσμα μη κυβερνητικών οργανώσεων και καλό είναι να μιλάμε μαζί τους γιατί πολλοί έχουν ε, πολλά και σημαντικά να προσφέρουν στο διάλογο. Η τρίτη ερώτηση ποια ήταν ένα λεπτάκι. Η προληπτική εποπτεία και ο επαρκής έλεγχος, μάλιστα. Δεν είμαι ε, σίγουρη αν μιλάτε για αυτό το είδος ελέγχων που μόλις σχολίασα. Ε, δηλαδή τους ελέγχους που διενήργησε η τράπεζα για την εκτίμηση των ε, μεσαζόντων και των άλλων ε, φορέων που προωθούν και υποστηρίζουν τα προγράμματα, τράπεζες και άλλοι δηλαδή, ή μιλάτε για τους ελέγχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ειδικού μας εξωτερικούς ελεγκτές ή την Εσωτερική Επιτροπή Ελέγχου. Για ποιους ελέγχους μιλάτε, μπορώ να σας πω περισσότερα αν θέλετε. Επόμενη ερώτηση. Ε, οι καταγγελίες, ε, γιατί αυξήθηκε, με ρωτάτε, ο αριθμός των καταγγελίων. Υποθέτω ότι αυτό μπορεί να αποδοθεί ε, στην καλύτερη γνώση των δραστηριοτήτων που είναι και αποτέλεσμα των εξηγήσεων που δίνουμε για ε, τα προγράμματά μας, για τη δραστηριότητά μας, για την προβολή που κάνουμε και όλοι ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε εμά ε, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λειτουργεί καλύτερο ο μηχανισμός καταγγελιών και έτσι έχουμε και περισσότερους πελάτες. Ε. Ε, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αυτό απηχεί μια αλλαγή επιτόπου. Νομίζω απλώ ότι είναι μια επιπρόσθετη ευκαιρία για να ακούμε τι πρόβλημα υπάρχει όταν υπάρχει. Τώρα σε σχέση με του χειρισμούς για την απάτη που έφτασαν στην ΕΤΕ για τι ε, χώρε ΑΚΕ που είναι και ε, ο τομέα που κατεξοχήν μα ενδιαφέρει από 6 σε 9 αυξήθηκαν οι καταγγελίε για να έχετε και μια εικόνα. Ε, όπως σας είπα όμως και στα εισαγωγικά μου σχόλια, ε, βλέπετε πώς οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι διαδικασίες έχουν αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό διότι Έχουμε τον αξιωματούχο για τα θέματα συμμόρφωση και το επιτελείο του αφενός που κάνει όλους ελέγχους για προληπτική εποπτεία, για την νομοθεσία, ε, για το ξέπλυμα χρημάτων, ε, για τις αντικρώμενες δικαιοδοσίες κτλ. Και από την άλλη έχουμε τον Γενικό Εισαγγελέα που ε, ερευνά όλες τις απάτε, όλες τι καταγγελίες. Πριν το 2005 δεν υπήρχε όλο αυτό το φάσμα, το πλωστάσιο στη διάθεσή μας. Ε, και που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτά τα ζητήματα ελέγχου. Μπορώ να σας δώσω και άλλα παραδείγματα, αν θέλετε να τα ακούσετε. Τώρα, μιλήσατε για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας. Μήπως... Ε, ε, με ενημερώνει ο συνάδελφος ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα μετά στη, στο επόμενο τμήμα που θα ασχοληθούμε με την έκθεση. Ούτως ή άλλως δεν είμαι ειδική γι' αυτό. Ε, ρωτήσατε αν θα υπήρξε αρνητική επίπτωση εντό ή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση με υποβάθμιση πιστοληπτική ικανότητα. Το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι συνειδητοποιούμε φυσικά την ε, ανάγκη και τη σημασία διατήρηση ε, τη βαθμολογία μα. Όπως πάντα, ε, χρειαζόμαστε να τηρήσουμε τα κριτήρια για τη, την κεφαλαιογική επάρκεια κτλ. Ε, ε, στα πλαίσια της εξωτερικής εντολής για τη χρηματοδότηση ευελπιστούμε ότι θα τηρήσουμε τα κριτήρια ε, Προ το παρόν διατηρούμε την ε, βαθμολογία μας ε, παρόλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρωζώνη, άρα παραμένουμε αισιόδοξοι για το μέλλον. Α, υπήρχε και μία ερώτηση για την για τον έλεγχο της τράπεζας. δεν κατάλαβα ακριβώς τι με ρωτήσατε. Ε, μιλάτε για μια συγκεκριμένη συμφωνία που έχουμε σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχουμε μια τριμερή συμφωνία. Ε, επειδή η ΕΤΕ είναι τράπεζα, είναι προφανές πως υπάγεται σε αυστήρα μέτρα ελέγχου, εξωτερικούς ελεγκτές, ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου, εσωτερικό ελεγκτικό τμήμα, οπότε δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιούσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα των φορολογούμενων, χρησιμοποιούσαμε με τόσο τακτικό και συστηματικό τρόπο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, νομίζω ότι γι' αυτό εξάλλου συνήθικε η συμφωνία με το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν την δυνατότητα συγγνώμη, να ελέγξουν κάποια από τα προγράμματα μας και ορισμένες φορές γίνεται αυτό και επιλέγουν όποιο πρόγραμμα θέλουν και το ελέγχουν. Αυτά για την εποπτεία. Άλλη δυνατότητα για την οποία ίσως ε, μιλήσατε όταν αναφερθήκατε στη μερική εποπτεία, ε, ίσως μιλούσατε για την, το μερικό έλεγχο του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Δεν είναι θέμα αυτό αρμοδιότητας μου. Νομίζω εσείς θα έπρεπε να απαντήσετε, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας διοχετεύσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται, ούτως ώστε να διεξαγάγετε και εσείς τους ελέγχους σας. Ε, οι μικροπιστώσεις ε, τώρα... υπάρχουν οι εκθέσεις στην επικαιρότητα ναι, για, για αυτό το θέμα. ξέρετε, ε, μιλάμε για μεγάλους αναπτυξιακούς κύκλους και όταν μιλάμε για μικροπιστώσεις ε, και βασιζόμαστε στην αρχή ότι χρειαζόμαστε άμεση δράση για να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Εξάλλου στο παρελθόν μικροπιστώσεις ήταν θέμα που διαχειριζόταν ο και χρειάζεται ε, διαρκώς να διοχετεύουμε στην αγορά κονδύλια και χρηματοδότηση ούτως ώστε να έχουμε μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ε, και οι πλέον φτωχοί ε, ρίψο κινδυνεύουν να ακολουθήσουμε μια εμπορική προσέγγιση να υπερχρεωθούν ε, κατά τη διαστολή. Εμείς θέλουμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα, το, τα τοκογλυφικά δάνεια και να προσθέσουμε κάτι σε αυτό το πλέγμα όσων ούτως ή άλλως χορηγούν τέτοια δάνεια στους φτωχούς, γιατί θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν σε στρεβλώσεις επί τόπου πάντως. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των μικροπιστώσεων εν γέννη είναι θετική για τους ε, μη έχοντες και κυρίως αυτοί που κινούνται πάνω από το όριο της φτώχειας ε, οι οποίοι, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούν να αποφεληθούν από αυτό το σύστημα, απλώ θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε επίπεδο συλλογικών αποταμιεύσεων ε, στις ντόπιε κοινότητε όπου ζουν. Πάντως, είναι πολύ θετική η εξέλιξη και είμαστε και περήφανοι για τη δική μας συνδρομή στην ανάπτυξη αυτών των θεσμών ε, χορήγησης ε, μικροπιστώσεων. Μπορώ να σας δώσω και άλλες λεπτομέρειες. Ε, αν όχι ακόμη σύντομα στην ιστοσελίδα μας θα έχουμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μικροδανείου για να δείτε ακριβώς ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της δράσης μας και έτσι νομίζω μπορώ να ολοκληρώσω και τον κατάλογο των ερωτήσεων αλλά όπως προείπα είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε και άλλες ερωτήσεις εδώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάρτον. Από την Επιτροπή υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, Το θέμα της αξιολόγησης του 3α αφορά γενικά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά ειδικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, δεν ακούω ερωτήσει. οπότε ευχαριστούμε ε, την ε, εκπρόσωπο και να δώσω τον λόγο ξανά στον κύριο Ρενχάζορ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την απάντηση στις ερωτήσεις μου. Βεβαίω. Φαντάζεστε πώς θα εξετάσουμε λεπτομερώς τις κατηγορίες που ακούστηκαν από την οργάνωση Counterbalance και το κάνουμε αυτό για να σας δώσουμε και την ευκαιρία να απαντήσετε και να ακουστεί αλήθεια. Δύο ερωτήματα τώρα που δεν απαντήθηκαν. Γνωρίζετε όλους τους τελικούς δικαιούχους των χρημάτων και έχετε ένα κατάλογο αυτών. Και δεύτερον, με αυτή την τριμερή συμφωνία υπάρχει η δυνατότητα το ελεγκτικό συνέδριο να συντάξει μια έκθεση για την, αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της απάτης μετά για τους συναδέλφους μου. Θα προσπαθήσω να έχω έτοιμο το σχέδιο έκθεσης μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, αλλά βεβαίως αν κάποιος επήγεται μπορεί να έρθει να με δει την ερχόμενη εβδομάδα και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. liebe ich Μάλιστα αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ και εγώ με τον εισηγητή, δηλαδή θα πρέπει να μπορέσουμε να θίξουμε αυτά τα ζητήματα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αυτό είναι μέρος του κοινοβουλευτικού ελέγχου μας και αυτό ήταν οι πολίτες από μας. Το ερώτημα τώρα το εάν μπορούμε να συζητάμε με μονομένες περιπτώσεις είναι ένα άλλο ερώτημα, αλλά οτιδήποτε σχετίζεται με διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω συμφωνούμε όλοι διακομματικά. Το δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε είναι κάτι το οποίο δεν απαντήθηκε ίσως αρκετά ξεκάθαρα σε ποιο βαθμό δηλαδή γνωρίζετε τους τελικούς δικαιούχους των χρημάτων αυτών. Ίσως μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα. Ε, μέσα στο μεγάλο κατάλογο έχασα αυτή την ερώτηση, είναι και από τις ευκολότερες. Βεβαίως πρέπει να έχουμε τον πλήρη κατάλογο των δικαιούχων όπου εμπλέκονται δάνεια της ΕΤΑ και έχουμε αρκετά στοιχεία για κάθε περίπτωση. Το θέμα για μας τίθεται ως εξής. Οι δικαιούχοι πρέπει να συμφωνήσουν για τη δημοσιοποίηση και πολλές φορές το δέχονται, γιατί από καιρού εις καιρών ρωτάμε κατά πόσο μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε τις υποθέσεις τους. Ίσως υπάρχουν και μερικές στο έγγραφο που σας έδωσα. Άρα ε, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει οι δικαιούχοι. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι υπό αυτή την έννοια έχουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από τα άλλα πιστοτικά ιδρύματα διεθνώς που πρέπει να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τους γιατί έχουμε την πιο απαιτητική πολιτική διαφάνεια, στο οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αποκαλύψουμε τα στοιχεία μας σε σχέση με τους δικαιούχους, υπό τον όρο ότι συμφωνούν οι δικαιούχοι. Αυτό ελπίζω να σας καθησυχάζει. Θα σας δώσουμε και άλλα στοιχεία, ε, αν το επιθυμείτε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Οπότε γνωρίζει η τράπεζα τους τελικούς δικαιούχους. Αλλά η δημοσιοποίηση απαιτεί και την συμφωνία τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάω τον λόγο. Ευχαριστούμε την κυρία Μπάρτον και την ομάδα της. Και νομίζω μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε στο επόμενο που επίσης αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ησυχητριά μας είναι η Ηλιάνα Ιβάνοβα, την οποία καλωσορίζω, όπως επίσης και τον κύριο Ντομινίκ Ντε Κρέανκουρ, Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Φένδυσεων. Να δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγήτρια, την κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ε, κύριε Ντεκρενκούρ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί συμμετέχετε, συμμετέχετε συγγνώμη, σε αυτή τη συνάντηση και γιατί ανταποκριθήκατε σε όλες τις συζητήσεις σε σχέση με την ΕΤΕ. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω το ρόλο της ΕΤΕ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα ήθελα να τονίσω τη, τα επιτεύγματα της τράπεζας το 2010 πριν ε, ε, κινηθώ στα ανησυχητικά ζητήματα. Βλέπουμε ότι ο στόχος των 30 δις έχει εκπληρωθεί για τις ΜΜΕ Επίσης ήταν η οδότηση για τις ΜΜΕ ε, και η εγκυοδοσία της τάξης του 2,8 δις, τα 60 δις επίσης και δόθηκαν 11 δις περισσότερα από αυτά που προβλέπονταν αρχικά. Επίσης αυτό αφορά και τις περιφέρειες σύγκλησης και θα ήθελα να σας συγχαρώ. Όμως τα βασικά ζητήματα που υπολείπονται έχουν ως εξής. Η βαθμολόγηση του τριπλού α, καταρχήν. Ορισμένα στοιχεία έχουν αλλάξει μετά από τη συζήτηση του Δεκεμβρίου. Είχαμε εξελίξεις ως προς τη βαθμολόγηση σε σχέση με το τριπλό α με αρνητικό outlook και πιστεύω ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να οριοθετήσει μια σαφή στρατηγική για μια σταθερότητα ως προς τη βαθμολόγηση και αν γίνει υποβάθμιση θα πρέπει να ξέρει τι οδό θα ακολουθήσει. Ως προς τις ΜΜΕ ως προς την υποστήριξή τους. Θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, καλύτερη λογοδοσία. Ιδιαίτερα αυτή η σύσταση αφορά τα μέσα της ΕΤΕ για τον έλεγχο των διαμεσολαβητών. Θα πρέπει να υπάρχουν benchmarks και ε, δείκτες διείσδυσης και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ανταποκρίνεται πλήρως η ΕΤΕ γιατί δεν είναι απόλυτα σαφές αυτό το πλαίσιο και αυτές οι ε, πληροφορίες για τους διαμεσολαβητές. Ένα άλλο θέμα είναι η εξωτερική δανειοδότηση της ΕΤΕ. Ε, συζητήσαμε για την ΕΤΑ Πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος της ε, δανειοδότησης, της ε, δανειοδοτικής δραστηριότητας και θεωρώ ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου που θα έπρεπε ε, για να αξιολογήσει την ΕΤΕ τη στιγμή που μιλάμε για κοινοτικά κονδύλια στα πλαίσια των εξωτερικών δραστηριοτήτων δανειοδότησης. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι ο κίνδυνος δανειοδότησης του συνολικού χαρτοφυλακίου. Εδώ μιλώ για το συνολικό επίπεδο πιστοτικού κινδύνου, επειδή υπάρχουν ε, μεγάλες πιέσεις λόγω της κρίσης, ε, της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Νομίζω θα πρέπει να καταπραίνουμε κάπως, να ελαφρύνουμε αυτό τον βασικό κίνδυνο. Ένα άλλο μάλλον ζητήματα που δεν είναι και τόσο σημαντικά αφορούν τα διαρθρωτικά ε, δάνεια. Τα προγράμματα διαρθρωτικών δανείων θα πρέπει η ΕΤΕ να παρέχει παρόμοια μέσα, αλλά όχι μόνο σε χώρες που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα και σε υγιείς χώρες και να μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για αυτά τα προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν να έχετε περισσότερα στοχοθετημένα προϊόντα για χώρες με καλή χρηματοπιστωτική πειθαρχία. Για το κατά πόσο θα ε, είναι μέτοχος της ΕΤΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα πρέπει να το δούμε και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να γίνει μέτοχος της ΕΤΕ το οποίο σημαίνει θα υπήρχε προωθημένη συνεργασία μεταξύ ΕΤΕ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, Υπάρχουν ε, δύο ζητήματα που θα ήθελα να θίξω και που δεν ε, αφορούν την έκθεση, αλλά πολλοί πολίτες ενδιαφέρονται και ανησυχούν σε σχέση με το θέμα της counterbalance που εφήγει στο πρώτο τμήμα το, της συζήτησης. Πρόκειται για μια υπόθεση στη Σερβία, στα, για νοσοκομεία της Σερβίας Πέρσι, στο τέλος του έτους, εστάλει μία επιστολή εξ ονόματος μίας σερβικής ΜΚΟ που έθιξε βασικά ζητήματα στην εφαρμογή ενός προγράμματος που χρηματοδότησε η ΕΤΕ. Ε, πρόκειτο για ανασυγκρότηση 20 ε, νοσοκομείων στη Σερβία με ε, δανειοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων το ίμιση θα καταβληθεί από την ΕΤΕ και το άλλο ίμιση από τη Σερβιγική Κυβέρνηση, από το Υπουργείο Υγείας και η επιστολή που ε, λάβαμε κάνει λόγο για καταχρήσεις, για κακή ποιότητα, κακή εφαρμογή, διαφθορά και έλλειψη αποτελεσμάτων καθώς και κακή εποπτεία των προγραμμάτων, του προγράμματος αυτού. Από όσο ξέρω υπήρξε κάποια επικοινωνία μεταξύ αρχών της ΕΤΕ και των αρχών που διερευνούν την υπόθεση και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την αξιοπιστία αυτών των δεδομένων, τι πρόοδος έχει επιτελεστεί και επίσης, ε, ε, από όσο γνωρίζω, υπάρχει και μία επικείμενη δραστηριότητα σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Σερβίας και εδώ εμπλέκεται ένα μεγαλύτερο ποσό, 200 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε Ποιε ποιες ε, ρήτρες διασφάλισης έχουν ληφθεί υπόψη έτσι ώστε να μην γίνουν καταχρήσεις εάν ανακύψουν με τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Μία άλλη υπόθεση που μας γνωστοποιήθηκε αφορά ένα πρόγραμμα στο Μαρόκο μιας γαλλικής εταιρείας η οποία ασχολείται με κέντρα αναψυχής σε εξωτικά σημεία. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση, η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΕ. Μιλάμε για 12 ε, εκατομμύρια μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού ποσού 75 εκατομμυρίων, αλλά δεν είναι σαφή σαφές κατά πόσο πραγματικά προωθήθηκαν οικονομικές δραστηριότητες επιτοπίως. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα έσοδα των, αυτών των κέντρων αψυχής και ξενοδοχειακών μονάδων και κατά πόσο τα κέρδη πάνε στους μετόχους. Δεν ξέρουμε λοιπόν ε, ε, κατά πόσο αυτή η εταιρεία που είναι μια μεγάλη επιχείρηση που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο ε, γιατί χρειάστηκε να χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕ. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια δηλαδή χρηματοδότησης για έγκριση παρόμοιων ε, projects. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ιβάνοβα. Θα ακούσουμε τώρα τις ομάδες και μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ποια θα ήθελε λοιπόν να μιλήσει. Λοιπόν, Κύριος Σκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σκιώδες μας εισηγήτρια δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Μου ζήτησε όμως να θέσω κάποια ερωτήματα για λογαριασμό της. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζει η ομάδα μας το σχέδιο έκθεσης και βεβαίως είναι διατεθειμένη να την παρακολουθήσει ε, επικοδομητικά. Τα τρία ερωτήματα τα οποία έχουμε είναι το εξή. Εμείς οπωσδήποτε θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όπως είχε απαιτηθεί και στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θέλαμε δε να υπενθυμίσουμε πως το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν μια νομική ανάλυση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Ανάλυση την οποία ακόμα δεν έχουμε λάβει και θα μας βοηθούσε στη δουλειά μας. Το δεύτερο ερώτημα απευθύνεται στην ΕΤΕΠ και μιλάμε για τα υπεράκτια χρηματοδοτικά κέντρα η δεσκιώδης εισηγητριά μας εδώ πέρα δεν βλέπει απέτηση από την ΕΤΕΠ να φροντίσει να μην οδηγεί η δραστηριότητα της ΕΤΕΠ σε φοροδιαφυγή ή και πλήσιμο ξέπλυμα χρήματος. Και κατόπιν Το ερώτημα το επόμενο είναι τα 3,2 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν δοθεί στην Ελλάδα ως δάνειο ε, σε σχέση με το κούρεμα το οποίο αναμένεται από στιγμή σε στιγμή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ, κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή και την εκπρόσωπο της ΕΤΕ κάτι για την υποστηρίξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συχνά συζητούμε το θέμα της υποστήριξης δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Στην παράγραφο 15 βλέπουμε 115.000 επιχειρήσεις ε, εποφελούνται από αυτή τη βοήθεια. Ο κ. Μπαρόζο στην ομιλία που έκανε την περασμένη εβδομάδα μας μίλησε για 24 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και είπε ότι αν κάθε επιχείρηση μπορούσε να προσλάβει έναν άνθρωπο, τότε θα λύναμε το θέμα της ανεργίας. Όταν κάποιοι από μας ε, συμμετείχαμε σε αυτή την ημέρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έγινε το φθινόπωρο. Ε, τουλάχιστον εγώ εκεί ήμουν. Υπήρχε μία πάγια καταγγελία ότι οι εκπρόσωποι ε, του επιχειρηματικού κόσμου στην Ευρώπη δεν ήξεραν καν πώς να χρηματοδοτηθούν. Θεωρούν ότι είναι πολύ περίπλοκο, υπερβολικά γραφειοκρατικό. Δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη των ταμείων και την ε, διαθεσιμότητα των κονδυλίων παρότι προβλεπόντουσαν για αυτές ακριβώς επιχειρήσεις. Ε, και αυτό το ακούγαμε μονίμως από όλους, τουλάχιστον εκεί στο σεμινάριο όπου συμμετείχα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι κάνετε από πλευρά σας. Είναι η ραχοκοκαλιά της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσει όπως σωστά έχει υποθεί. Άλλη ερώτηση τώρα για την παράγραφο 48. Η e Η ΕΤΕ λέει εδώ ότι δεν θα έπρεπε να υποστηρίζει οτιδήποτε βλάπτει το κλίμα. Αυτό δηλαδή καλύπτει και τους αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, ότι βλάπτει το περιβάλλον. Τι νοούμε. Ε, ούτε την πυρηνική ενέργεια μπορεί να υποστηρίξει μέσα από τα προγράμματα. Είμαι περίεργος ε, να, καταλάβω, διότι στην Ευρώπη, λένε και περισσότερο, βασιζόμαστε στο φυσικό αέριο της Ρωσίας. Το πετρέλαιο που νομίζουμε θα το βρούμε δεν ξέρω, αλλά πάντως ε, προβλήματα έχουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σμιτ. Κυρία Χολμάια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν σε άλλη επιτροπή, οπότε θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση σε ένα άλλο θέμα στο θέμα 4. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις απαντήσεις που έδωσε και το ερώτημα είναι το εξής. υπάρχει μία ομάδα παρακολούθησης η οποία συστάθηκε ακριβώς για να μπορεί να διαπιστώσει το εάν επιτυγχάνονται οι στόχοι της αναπτυξιακής βοήθειας, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, ποια προβλήματα προκύπτουν και το ερώτημα είναι αν στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μάλιστα. Ένας ακόμα συνάδελφος, ο κύριος Μπαλτσίτης, αν οι υπόλοιπε ομάδες δεν θέλουν ε, να τοποθετηθούν, τότε να ακούσουμε τον κύριο Παλτσίτης. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση. Η ΕΤΕ εξακολουθεί να έχει την ανώτατη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας. Γίνονται πολλές συζητήσεις ε, για την ε, βαθμολογία και υποβαθμίστηκε κατά τι ε, η βαθμολογία σας και λένε κάποιοι ότι πρέπει να κάνετε τα πάντα ούτως ώστε να αναβαθμιστείτε και πάλι. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας άποψη και το μέλλον πώς, στο μέλλον πώς θα τοποθετηθείτε διότι εδώ στο Κοινοβούλιο αρχίζουμε να συζητάμε για την δυνατότητα σύστασης ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης. Μάλιστα. Νομίζω μπορούμε να απαντήσουμε αυτά και να περάσουμε μετά σε ένα δεύτερο γύρο. Όχι, όχι. Εγώ προτείνω να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Γιατί ακούστηκαν αρκετά. Οπότε θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ντεϊκρή Γιανκούρ. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχίζοντας... Ε, Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την τόσο καλή έκθεση και για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Καθ' όλη την ε, ε, διάρκεια της διαδικασίας διάθεσης πληροφοριών, διαλόγου για το έργο μας Νομίζω ότι πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνειδητοποιήσει ότι ακολουθεί ε, κατά πόδα στις συστάσεις ε, του Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα ε, να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία-τέσσερα σημεία μόνο, όχι ισχυριζόμενο ότι είναι τα βασικότερα σημεία αυτή, αλλά ε, κρίνω ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν παρανοήσει ή αξίζει να συζητηθούν απλώ. Πρώτον, ε, και δεν τα λέω, δεν το αναφέρω κατά σειρά προτεραιότητα. Ακολουθώ τη σειρά την οποία έχουν στην έκθεση. Πρώτο λοιπόν το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όντω, η έκθεση αναγνωρίζει τις ε, προσπάθειες ε, που έχουν γίνει και τα επιτεύγματα της Τράπεζας για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεσούσης της κρίσης. Ε, το τμήμα αυτό της ε, Τράπεζας ε, και τα εταιρικά κονδύλια που εγκρίθηκαν εσχάτως αναδεικνύουν σε προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 2012 θα αυξηθούν την περαιτέρω τα κονδύλια σχέση με προηγούμενα έτη ε, δεδομένου του ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν συρρυκνωθεί τα κονδύλια χρηματοδότηση, αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Επίσης, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζουμε κοινά εργαλεία για να εκμεταλλευτούμε την μόχλευση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εκεί εντάσσεται και η επιχείρησή μας στην Ελλάδα, καθώς επίσης ε, και ε, ε, ο μηχανισμός διευκόλυνσης της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καταμερισμό του κινδύνου. Ε, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ε, των μεσαζόντων. Δεν θα επεκταθώ για αυτό το θέμα, εκτός αν μου το ζητήσετε. Μπορώ πάντως ε, να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν τα στοιχεία στην ιστοσελίδα. Υπάρχει μια διαφανέστατη παρουσίαση της μεθόδου επιλογής των μεσαζόντων. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που έχουν ιδιαίτερο βάρος για την επιλογή τους. Πρώτον, είναι το κριτήριο της προσθετικότητας, ε, δηλαδή θέλουμε όχι μόνο να αναχρηματοδοτούμε τις ε, τράπεζες, και αυτό σημαντικό βέβαια είναι, αλλά θέλουμε να δίνουμε περισσότερα κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ε, άλλο κριτήριο, ποιο είναι το οικονομικό όφελος που προσφέρουμε και αν αυτό μετακυλίεται στον τελικό δικαιούχο και δεν σταματάει κάπου σε αυτή την αλυσίδα μεσαζόντων τρίτων. Ε, να απαντήσω στην ερώτηση του κύριου Σμιτ, αν θυμάμαι καλά, το θέμα δηλαδή της διαφάνειας, η υποχρέωση, δηλαδή συμβατική υποχρέωση, να ενημερώνουν ε, οι μεσάζοντες ε, τους τελικούς δικαιούς της μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΤΕ. Η έλεγχη είναι μια άλλη διάσταση αυτού του ίδιου ζητήματος των μικρομεσαίων Φυσικά έχουμε εκτεταμένους ελέγχους επιτόπου, ε, προβλέπονται ελέγχει και φυσικά αυτό που θέλουμε είναι να αποζημιωθούμε όταν χορηγούμε ένα δάνειο. Άρα έχουμε κάθε συμφέρον να εποπτεύουμε μαζί με τους μεσάζοντες την κατάσταση και να βλέπουμε κατά πόσο ε, ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ε, οι δικαιούχοι. Τώρα για την υποβολή εκθέσεων και συγκεκριμένα προς το Κοινοβούλιο ε, σας διαβεβαιώ ότι καταγράψαμε όλα τα αιτήματά σας Επίσης, αν υπάρχουν ad hoc ερωτήσεις, μην διστάσετε διότι ε, με συστηματικό τρόπο διοικητεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάφορες εκθέσεις και ενημερωτικά σημειώματα. Πιστεύω ότι είστε ικανοποιημένοι με, τις με την ενημέρωση που σας ε, παρέχουμε. Εάν όχι, ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τη μέθοδό μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα αναρωτιόμαστε τι μέτρα θα μπορούσαν να αναλυθούν εν ώψη και της επικείμενης Ευρωπαϊκής Συνόδου στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Πιστεύω ότι θα είναι ύψιστη προτεραιότητα στη μέση διάταξη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και όλα τα υπόλοιπα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότησή τους, από κοινού δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την δράση της ΕΤΕ. Τώρα, ε, για την εποπτεία και τους ελέγχους θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Αρχίζοντας να πω ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση ανάμεσα στα δύο. Πρώτα απ' όλα. Το υπάρχει το θέμα του οικονομικού ελέγχου auditing, όπου η σωστή επαλήθευση του κατά πόσο οι δραστηριότητες της τράπεζας υπάγονται στους κανόνες και τα ε, πρότυπα ε, που έχουμε και τις πρακτικές που πρέπει να τηρήσουμε για αυτού του είδους του ελέγχους λοιπόν έχουμε ολόκληρο οπλοστάσιο μέσων. Ε, εσωτερικός έλεγχος, ο γενικός ελεγκτής της τράπεζας, εξωτερικοί έλεγκτες, εσωτερική επιτροπή ελέγχου και, και ούτω καθεξής. Ε, από πλευράς λοιπόν οικονομικού ελέγχου, οι κανόνες ε, του παιχνιδιού είναι τέτοιοι ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων μας. Ε, δεύτερον, έχουμε το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου και θέλω να το τονίσω αυτό, διότι αναφέρθηκε, ε, είναι ξεκάθαρο κάθαρο ηλίου φαϊνότρων ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει κάθε δικαίωμα να ελέγξει η αδίποτε δραστηριότητα της τράπεζας που χρησιμοποιεί κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης. Αυτό είναι συμπεφωνημένο, ε, είναι βίβλος, ε, καταγράφεται και στην τριμερή συμφωνία με την Επιτροπή και το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αμφιβολία δηλαδή για αυτό το θέμα. Ε, και ήδη έχουν ε, υποβληθεί αιτήσει ε, για περαιτέρω ελέγχου που συνάδουν απολύτω και με το πνεύμα διαφάνεια που χαρακτηρίζει την εταιρεία. Στο σημείο 3 της έκθεσης για τη Βασιλεία 3 Ε, δεν νομίζω ότι τίθε κάποιο θέμα διαφορετικό σε σχέση δηλαδή με τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μεταγραφούν αυτά στην νομοθεσία της Ένωσης θα τα υλοποιήσουμε, αλλά ούτε καν περιμένουμε ε, για να εφαρμόσουμε δηλαδή τις προθέσεις της Βασιλείας 3 στο δικό μας έργο. Αυτό σχετίζεται με την κεφαλουχική επάρκεια για υποστήριξη των δραστηριοτήτων, κανόνες για τη ρευστότητα, δεν θα σας κουράσω τώρα με τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα το πνεύμα της Βασιλείας Τρία το τηρούμε ακόμη και πριν ε, ενσωματωθεί στην νομοθεσία ε, της ε, Ένωσης. Ο κύριος Γκέγερ με ρώτησε κάποια πράγματα για την παρακολούθηση η ΕΤΕ είναι απολύτως διαφανής, νομίζω το γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε. Κανένας ε, πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός, ούτε κανένας εθνικός οργανισμός υπάγεται σε ένα τέτοιο έλεγχο, σε τέτοια παρακολούθηση όπως η ΕΤΕ. Παρόλα αυτά, ξέρετε, δεν μας ενοχλεί αν είναι να λειτουργήσουμε ως παράδειγμα, ως πρότυπο, αν είμαστε προτεργάτες, αν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν ε, και ε, ο οργανισμός που θα μπορούσε να το εφαρμόσει αυτό είναι η ΕΚΤΕ λόγω του θεσμικού της ρόλου αλλά τα κράτη-μέλη δεν τον έχουν δεχτεί. Ο πρόεδρος ε, της ΕΚΤΕ αναφέρει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει πλειοψηφία προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, τώρα η EBA παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να μας βοηθήσει αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί πλήρης έλεγχος. Εμείς συνεχίζουμε να λειτουργούμε παρά τις εποπτείες ε, και σε συνεργασία με την ε, Λουξεμβουργιανή Εποπτική Αρχή συνεχίζουμε να λειτουργούμε χωρίς να έχει βρεθεί ακόμη ικανοποιητική νομική λύση σε σχέση με τους οικονομικούς ελέγχους. Θέλω να γίνει διάκριση με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση, monitoring and evaluation, διότι ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι των προγραμμάτων και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ευθυγραμμίζονται με τους αρχικούς στόχους. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσω απαντώντας έτσι και στην ερώτηση της κυρίας Χολ ότι η οργάνωση της τράπεζας για την παρακολούθηση ενισχύθηκε πρόσφατα και από την αρχή του 2012 πλέον ε, έχουμε ένα νέο σύστημα ε, μέτρησης, καταμέτρησης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ε, και το αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας ε, θα υποβληθούν στο ε, Κοινοβούλιο εφ' και ελπίζω έτσι να καλύψουμε τις προσδοκίες που έχετε για αυτό το θέμα. Τρίτον, τα ορυκτά καύσιμα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα αριθμητικά στοιχεία. Σε ένα σχέδιο έκθεση από την Επιτροπή Περιβάλλοντο υπάρχει ένα αριθμητικό στοιχείο που είναι πλημελέ, ε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Φυσικά δεν δίνουμε 10% των δανείων για ορυκτά καύσιμα. Πόρο απέχουμε από ένα τέτοιο ποσοστό. Το πραγματικό ποσοστό ε, είναι 3,5% περίπου. Ε, της δανειοδοτικής μας ικανότητας ε, για την ε, παραγωγή, για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και περνάμε από το λιγνίτη, από μονάδες μάλλον για άνθρακα και λιγνίτη. 66 100% της δανειοδότησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διοχετεύονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία λεπτομερή ως συνήθως. Παρακαλώ προσοχή όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα μεγέθη. Γιατί έχουμε ακόμη δραστηριότητες ε, υπέρ της εκμετάλλευσης ορεικτών καυσίμων. Ε, λοιπόν, όπως είπε σωστά και ο κύριος Σμιτ, για τους προφανείς ε, λόγους, δηλαδή ότι υπάρχει και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, της τροφοδοσίας, της ένωσης δεν μπορούμε ακόμη να καλύψουμε τα πάντα από τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, ε, κυρίω σε κάποιες μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, Φερρυπίν, ε, που αποφάσισαν να ε, σταματήσουν την παραγωγή πυρηνική ενέργειας. Το φυσικό αέριο, παραδείγματο χάρη, ακόμη χρήζει χρηματοδότησης, παρότι μόνο οριακά στην περίπτωση τη ΕΤΕ, Έχουμε πολύ αυστηρούς λοιπόν περιορισμούς και το ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 3,5% για την δανειοδότηση για την παραγωγή ε, ηλεκτρικής ενέργειας, άνθρακας και λιγνίτης. Οι όροι υπάρχουν, είναι διαθέσιμοι, είναι τεχνικοί οι όροι, δεν χρειάζεται το να σας κουράσω. Ε, πάντως είναι ιδιαίτερα αυστηρή έλεγχη και συγκεκριμένοι περιορισμοί και κυρίως τίποτα δεν αναλαμβάνεται όταν αντιβαίνει στους γενικότερους στόχους ένωση για τη μείωση των εκπομπών και για την προστασία του περιβάλλοντος το άνοιγμα σε όλες τις χώρες ε, για τις δραστηριότητες της ΕΤΕ είναι ένα θέμα που σχολίασε κάποιος από όλους. Κοιτάξτε, χθες στην Επιτροπή Ρέτζη είπα το εξή. Αν δεν υπάρξουν μέτρα συγκεκριμένα για τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε μέτρα που να ισχύουν για όλες τις χώρες, να μην επιβάλλουμε περιορισμούς στα υφιστάμενα μέτρα. Αυτή είναι η άποψή μας. Ε, για το τριπλό α τώρα, γιατί είναι ένα θέμα που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Ε, στα τέλη του 2011 αυτό το θέμα του τριπλού α της ΕΤΕ προέκυψε, αν θέλετε, ε, ε, στον απόϊχο της συνολικότερης συζήτησης για την πιστοληπτική ικανότητα όλων των χωρών της ε, Ευρωζώνης. Η Standards and Poor's ήταν η πρώτη που μας έθεσε υπό υποπτία, γι' αυτό το λόγο και ανακαλύψαμε και παρεμπιπτόντως μα δημιουργεί δυσκολία αυτό. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι οι οίκοι αξιολόγηση έχουν τροποποιήσει την προσέγγιση που ακολουθούν και τη μέθοδο που χρησιμοποιούν ε, προ ανάλυση ε, της πιστοληπτικής ικανότητας. Στο παρελθόν ε, επικεντρώνονταν ω επιτοπλήγων στην κεφαλουχική επάρκεια, δηλαδή ε, πόσα κεφάλαια έχει η τράπεζα σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού κινδύνου και άλλαξε αυτό λοιπόν πρόσφατα χωρί να ενημερωθούμε κατά το δέον και πέρασαν σε ένα άλλο δείκτη, τη μόχλευση. Ποια είναι η μόχλευση, ε, ονομαστικός λόγος ε, ε, του συνόλου των δανείων ε, προς ε, των συνολικών κονδυλίων. Και είχαμε πολύ ψηλότερη μόχλευση σε σχέση με άλλες πολυμερές τράπεζες για τον απλό λόγο ότι κατά 90% εμείς δραστηριοποιούμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχυρότερες χώρες μεγαλύτερο κίνδυνο και αυτό μας επιτρέπει ε, με ονομαστικούς όρους να έχουμε μειωμένο κεφάλαιο σε σχέση με άλλες ε, ε, τράπεζες. Έχουμε λοιπόν υψηλό δίκτυο μόχλευση και γι' αυτό το λόγο μας έδεισαν υπό υποπτία. Ε, συζητήσαμε στο τέλος του 2011 με τους διάφορους οίκους αξιολόγησης, ε, ήρθαν και εξέτασαν εξονυχιστικά το χαρτοφυλάκιό μας και δέχτηκαν ότι και εκείνοι οι ίδιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν το τριπλό α, άρα ήραν αυτή τη διαδικασία εποπτείας ε, και λόγω της χάρη στην ποιότητα του χαρτοφυλάκιου αποκατέστησαν το τριπλό α, αλλά παρόλα αυτά παραμείναμε υπό δυσίωνες οικονομικές ε, προοπτικές. Ε, παρά την υποβάθμιση των μετόχων και μέρους ε, πιστωτών μας, έτσι, βάσει του χαρτοφυλακίου, χάρη στην ποιότητα αυτού του χαρτοφυλακίου καταφέρουμε να διατηρήσουμε την επιστοληπτική ικανότητα, μειώνοντας ε, το συνολικό όγκο δανείων και κατεβάζοντας το λόγο της ε, μόχλευσης κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, τέθη το ζήτημα του κουρέματος, απομείωσης ε, του δανείου που συζητάμε για την Ελλάδα, θα ήθελα ε, ε, πολύ απλά να σας πω εδώ ότι πιστεύουμε και πραγματικά είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Αν υπήρχε κάποια ιδέα να εφαρμοστεί αυτό το ε, αυτή η απομείωση της ΕΤΕ, αυτό ε, θα κατέλειε πάρα αυτά το τριπλό α. Ε, δεν είμαστε ΕΚ, δεν βγάζουμε χρήματα, δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουμε προϋπολογισμό. Εμείς ζούμε από τα δάνεια της αγοράς. 400 δις ομολογιών έχουμε στις αγορές ε, και νομίζω ότι είναι γενικώ αποδεκτό ότι ε, έχουμε ένα ευμενές καθεστώς ε, για την πιστοληψία και έτσι λειτουργούμε γιατί αλλιώς ε, τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία της τράπεζας. 70% περίπου ε, των δανείων μας βασίζονται σε οργανισμούς που λόγω των δικών τους ε, κανόνων υποχρεούνται να αγοράζουν ομολογίες τριπλού α. Αν χάσουμε εμείς το τριπλό α, στη δική μας ε, ιδιάζουσα περίπτωση. Αυτό θα θέσει να αμφιβόλο ε, την ίδια την υπόσταση και τη λειτουργία τη ε, τράπεζα. Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε το τριπλό α, επιβεβαιώθηκε το τριπλό Α λόγω τη ποιότητα ε, του χαρτοφυλακίου μα, για να ανακεφαλαιώσω. Δεν περιμένουμε να συμμετάσχουμε καθιονδήποτε τρόπο στο PSI για την Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε φυσικώς να βοηθούμε την Ελλάδα. Αν αλλάξει κάτι ε, σε αυτές τις αποφάσεις ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα λεπτό για την τράπεζα. Θα ήθελα να κάνω μία σύντομη αναφορά, επιτρέψτε μου, για αυτά τα δύο προγράμματα στα οποία αναφέρθηκε η συγγήτρια για το θέμα των ε, νοσοκομείων στην ε, Σερβία. Δεν μπορώ να το σχολιάσω περαιτέρω, μπορώ να σας πω μόνο ότι διεξάγεται τώρα η έρευνα εις πλήρη γνώση της Όλαφ και, ε, γνώση της Όλαφ και όταν περατωθεί ο έλεγχος θα σας διαβιβάσουμε τα πορίσματα, προς το παρόν δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ε, και κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου και δικαίω. Έχουμε πελήρη αντίληψη της κατάστασης, θα επανέλθουμε. Ε, για το θέμα του Μαρόκου, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δουν ε, ένα, μια απάντηση είναι ερωτηματολογίου σε όλες αυτές τις καταγγελίες της counterbalance. Λοιπόν, ε, ανησυχεί η τράπεζα σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την χρήση αυτών των επιχείων τίτλων από πλευράς ε, της counterbalance αντί να υποστηρίζουν ε, τους λόγους για τους οποίους χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή για να ε, Ξηθεί ενημέρωση σε σχέση με τα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Το αντίθετο κάνουν. Συστηματικά υπονομεύουν το έργο μα με πλημελείς ισχυρισμού και καταγγελίε και μα ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό το φαινόμενο. Έχουμε ε, τα δεδομένα, έχουμε τα στοιχεία, είναι στη διάθεσή σας. Πρόκειται για ένα τουριστικό πρόγραμμα. Ο τουρισμό είναι σημαντικότατο τομέα στο Μαρόκο ε, και πολλοί ντόπιοι απασχολούνται σε αυτό το τομέα. Αυξήθηκε η απασχόληση, το θέμα του περιβαλλοντικού, κοιτάξτε, εξετάσαμε διεξοδικά και αυτή η εταιρεία που προωθεί το πρόγραμμα είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ως προς ε, την γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Υπάρχουν ε, όλα αυτά τα στοιχεία διαθέσιμα. Δεν θέλω να ε, σπαταλώ το χρόνο σας με αυτά. Είναι στη διάθεσή σας και μπορούμε να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Äh, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναλυτικές σας απαντήσεις. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρω. Ο κύριος Κάλβιν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της τράπεζας και να συγχαρώ και την ε, συντάκτη της έκθεσης. Ένα ζήτημα θα ήθελα να αναφέρω μετά από τα σχόλια του προσώπου της τράπεζας αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτήν. Εμείς πιέζουμε συνεχώς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, για να στηρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα είναι μια τράπεζα. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Και όταν αρχίζουμε να κάνουμε ερωτήσεις για την αξιολόγηση μιας τράπεζας, πρέπει να είναι σαφές ότι καμιά στιγμή, κάποια στιγμή οι απαιτήσει του Κοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων μπορεί να είναι αντιφατικές με τις απόψεις των οίκων αξιολόγησης. Όταν λοιπόν λαμβάνουμε αποφάσεις πρέπει να αποφασίζουμε τι είναι πρώτη προτεραιότητα. Και θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο αναφέρει εδώ πέρα η κυρία Ιβάνοβα, αυτό το οποίο προτείνεται, ότι στην περίπτωση αυτή η ε, αξιολόγηση μπορεί να είναι η κορυφαία προτεραιότητα, γιατί αν για τον οποιονδήποτε λόγο χάσει την αξιολόγηση αυτή θα ε, χειροτερεύσουν τα πράγματα και ως προς τους στόχους που έχει. Οπότε ως προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτή η πρώτη και να συνεργαστούμε με την τράπεζα για να διατηρηθεί το 3α είναι πολύ θετικό το ότι μας εξήγησε ο κ. Ντεκονκού τον λόγο των ε, πρόσφατων ερωτήσεων για τις αξιολογήσεις και τη μεθοδολογία της τράπεζας και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε την αξιολόγηση μαζί με το σχέδιο της τράπεζας είναι να αναζητήσουμε τρόπους να δώσουμε όχι περισσότερο κεφάλαιο αλλά περισσότερα μετρητά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί το να αλλάξει η προσέγγιση ε, των οίκων επενδύσεων από την κεφαλαϊκή επάρκεια στη μόχλευση ε, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω, μέσω του να αυξήσουμε τα μετρητά της τράπεζας. Οπότε, όταν θα συζητάμε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα μπορούσαμε τότε να εξετάσουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα μετρητά που υπάρχουν στη διάθεση της τράπεζας και πάλι στην έκθεση υπάρχει μια πρόταση η οποία έχει ε, επαναλάβει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο δηλαδή να διασφαλιστεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κεφάλαιο της τράπεζας. Όχι μορφή εγγύησεων, αλλά υπομορφήν ρευστού. Και με αυτό τον τρόπο, σε συνδυασμό ε, νομίζω με τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το μετρητό που υπάρχει στη διάθεση της τράπεζας. Σας ευχαριστώ. Γιάνν Γκερμπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της τράπεζας για τις απαντήσεις του στον πρώτο γύρο κρίσιμη σημασία για εμάς είναι να υπάρχει μια συνέπεια στην ε, πολιτική μας. Όχι αντιφατικότητα. Αυτό βέβαια στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε πως κάποιες πολιτικές είναι πιο ίσες από τις άλλες ε, που έλεγε και ο συγγραφέας. και φαίνεται πως μία από τις πολιτικές της λιγότερο ίσως είναι η βιοπικιλότητα. Υπήρχε μια στρατηγική μέχρι το 2010 που έλεγε πως θέλαμε να σταματήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας, τώρα έχουμε μια νέα στρατηγική και πάλι το 2020 θέλουμε να σταματήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας και αποκατάσταση το ερώτημά μου είναι με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακολουθεί τους στόχους αυτούς στα έργα της. Υπάρχουν ιδέες περί μιας αρχής μη απώλειας, δηλαδή αναέργο να μην υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στη βιοπικιλότητα και αν υπάρχει να αντισταθμιστεί κάπου αλλού. Αυτό βεβαίως ε, είναι κρίσιμο για τους στόχους ε, αυτούς και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους λέμε τη φύση ασφάλεια ζωής. Ε, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικός τομέας, αλλά έχει εξαιρετική σημασία θα μπορούσατε ίσως ε, να μας πείτε κάποια πράγματα από αυτό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσέσκοβα, παρακαλώ. Ε, <clears throat> ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτριά μας καθώς και την εκπρόσωπο της ΕΤΕ για όλες τις πληροφορίες οι οποίες είναι άκρος ενδιαφέρουσες σε σχέση και με τις επιλογές που διανοίγονται για την ΕΤΕ δηλαδή την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Από ό,τι καταλαβαίνω, η ΕΤΕ δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης. Τώρα με βάση τις συζητήσεις πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανεξαρτησία της ΕΤΕ. έτσι ώστε η τράπεζα να κρατήσει τη θέση της, να εδραιώσει τη θέση της στις, στις αγορές κεφαλαίων. Γι' αυτό έγινε λόγος και για τους ε, ενδιάμεσους μηχανισμούς, τους μηχανισμούς γενικότερα, για να μην υπάρχει αναστολή δραστηριοτήτων της ΕΤΕ. Τώρα, ως προς τις ε, ΜΜΕ και την υποστήριξή τους, ιδιαίτερα εντός ε, Ένωσης, Διαβάσαμε την έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου, το συζητήσαμε στην Επιτροπή μας τη Δευτέρα και μάθαμε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους και την εποπτική διαδικασία των δανειοδοτήσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να θίξω το εξής ζήτημα. Θα ήταν δυνατόν η ΕΤΕ να ελέγξει την κατάσταση των τελικών δικαιούχων. Δηλαδή πώς χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους οι δικαιούχοι. Γιατί ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της έκθεσης είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος των νέων θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εξαιτίας ε, μάλλον χάριν αυτών των δανείων. Δεν ελέγχονται οι θέσεις απασχόλησης. Αυτό το οθήγω ως παράδειγμα σε σχέση με τη θέση των δικαιούχων. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο, οπότε θα ήθελα να ζητήσω ξανά από τον εκπρόσωπο της τράπεζας να απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Εντάχη, προς τον κύριο Κάλφιν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τα όσα προανέφερε. Νομίζω ότι το θέμα αυτή τη στιγμή για την ΕΤΕ είναι να δώσει μεγάλη μάχη και να θέσει οροφές ε, ως προς τη δραστηριότητά της ως προς τις ε, κεφαλαιακές ροές και συνεπώς θα πρέπει να ενισχύσουμε τον παρονομαστή έτσι ώστε να έχουμε ε, μία διαδικασία μόχλευσης για τον αριθμητή της τάξης του 7. Δηλαδή κατά πόσο το 1 ευρώ μπορεί να μετατραπεί σε 7 ευρώ με βάση τον ε, δίκτυ μόχλευσης της τράπεζας. Δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε μία σχέση ένα προς 7. Προς κύριο Γκαμπάντη θα ήθελα να πω ότι δεν έχω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι η ΕΤΕ σκέφτεται πολύ σοβαρά αυτό το θέμα της βιοπικιλότητας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους που ασχολούνται με κάθε επιμέρους τομέα και προβλέπουμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την βιοπικιλότητα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε μπορώ να σας φέρω σε επαφή με τους υπευθύνου. Ως προς τις ΜΜΕ, το τρίτο θέμα που θίξατε γνωρίζετε ότι απασχολούμε 1.800 άτομα προσωπικό, ε, όλοι σχεδόν βρίσκονται στο Λουξεμβούργο. Και αν θέλουμε να υπάρχει μια διάδραση με τις 150.000 ΜΜΕ, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα παρά τους ε, διαμεσολαβητές. Αυτό αφορά και αυτά που είπε η κυρία Τσεσακόβα σε σχέση δηλαδή με τον έλεγχο των μεμονωμένων ΜΜΕ και τον έλεγχό τους. Φυσικά δεν κάνουμε ό,τι θέλουν. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια σαφή μελέτη και περιγραφή για το τι είναι δυνατό, τι δεν είναι δυνατό, τι είναι επιλέξιμο και ούτω καθεξής. Και οι τράπεζες διαμεσολαβητές θα πρέπει να τα ελέγξουν αυτά. Εμείς ως ΕΤΕ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, δεν θα ήταν εφικτό. Θα ήθελα να προσθέσω ότι το θέμα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι φαίνεται αρχικά. Ορισμένες επενδύσεις δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας, άλλες δημιουργούν καινοτομία με λιγότερες θέσεις αλλά με καλύτερο μέλλον. Άρα θα πρέπει να το δούμε συνεκτικά. Δηλαδή δεν μιλάμε για το πόσες θέσεις δημιουργεί κάθε ΜΜΕ ξεχωριστά. Δεν θα ήταν ε, σωστή αυτή η αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ορίσουμε την επιλεξιμότητα μίας ΜΜΕ από τις θέσεις και μόνο εργασίας που δημιουργεί. Θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία που θα δημιουργήσει αργότερα θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Διευθυντά για τις απαντήσεις σας. Τώρα τον λόγο έχει η συγκήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους, τις παρεμβάσεις τους. Καλώς ορίζω επίσης ε, τις ε, απαντήσεις του κυρίου Ντεκρινικούρ. Καλώς ορίζω ιδιαίτερα την ειλικρίνεια και την διάθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο για το κομμάτι εκείνο που ε, βεβαίως είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτό περισσότερο ήταν πρόσκληση στο ελεγκτικό συνέδριο παρά προς εσάς. Τώρα για τα συγκεκριμένα σχόλια των ομάδων από τις ε, πολιτικές ομάδες για τους σοσιαλδημοκράτες συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκαΐρ για τα offshore και το 3α τις υπεράκτες εταιρείες. Πράγματι τα έχω στην και σε ευχαριστώ. Το σχόλιο του κυρίου Σμιτ και κάποιοι συναδελφοί ανέφεραν το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικό και έχει θέση στην εκθεσή μου ως ε, υπότιτλος αν θέλετε για την εντολή εσωτερικού δανεισμού της τράπεζας. Τώρα για την παράγραφο 48 το θέμα που αφορά την κλιματική αλλαγή ε, εγώ δεν βλέπω ε, αναφορά σε σταμάτημα χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων. Αυτό το οποίο ζητάω είναι τα έργα να συμμορφώνονται με αυτά τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική. Αυτό. Τώρα, σημείωσα αυτό το οποίο είπατε κύριε Ντεκριανκούρ για τα στοιχεία περιορυκτών καυσίμων. Αυτά μου τα έδωσαν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν τα έλεγξα, αλλά ευχαρίστως να το δω και να τα διορθώσω. Πέρα από αυτά, νομίζω πως όλα τα υπόλοιπα είναι σαφή. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων και ελπίζω και η έκθεση να σας βοηθήσει στο μέλλον. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε... Ευχαριστούμε την κυρία Ιβάνοβα και τον κύριο Ντεκραγενκούρ. Τελειώνει και το σημείο 4 και περνάμε στο επόμενο, το 5. Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας του Όλαφ. Η Ίγκεμποργ Γκρέσλε είναι η εισηγήτρια και εδώ πέρα καλωσορίζω την Ρόζαλιντ Ράιτ και την... Ε, το μου εδώ πέρα, ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής. Θα παρουσιάσετε λοιπόν την έκθεση και καλωσορίζω βεβαίως και τον Γενικό Διευθυντή του Όλαφ, τον κύριο Τζοβάνι Κέσλερ. Η εισηγήτρια θα ήθελε να κάνει κάποια εισαγωγή. Όχι. Να περάσουμε κατευθείαν λοιπόν στην έκθεση. Να παρακαλέσω λοιπόν την κυρία Τεάτο ε, και τις δύο εισηγήτρες να ξεκινήσουν. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Κυρία Τεάτο. Danke. Ähm, Herr Präsident, äh, sehr geehrte Frau Berichterstatterin, meine Damen und Herren Abgeordnete. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ εγώ και η συνάδελφός μου για το ότι έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την έκθεση δραστηριότητας της Επιτροπής μας. Είναι η τελευταία μας έκθεση για τη λίγη δική μας θητεία και τα νέα μέλη ούτως ή άλλως έχουν ξεκινήσει τη δουλειά τους. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκθέσεις μας, αυτή τη φορά δεν περιγράφουμε μόνο τις δραστηριότητές μας το 2011, αλλά παρουσιάζουμε και τη δουλειά μας τα προηγούμενα έξι έτη. Η βασική έκθεση λοιπόν της εντολής μας ήταν να ελέγξουμε την ανεξαρτησία του Όλαφ χωρίς να μπούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η εποπτεία του Όλαφ λοιπόν επικεντρώθηκε σε τρεις σημαντικούς τομείς. Πρώτον, στην εφαρμογή της ερευνητικής λειτουργίας του Όλαφ. Δεύτερον, στις επιπτώσεις της διαχείρισης του Όλαφ στην ανεξάρτητη αυτή λειτουργία και τρίτον στην εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων ως εγγύηση της ανεξαρτησίας του Όλαφ. Στη σημερινή μας παρουσίαση έχουμε κάνει μια επιλογή των σημαντικότερων πτυχών για τα ζητήματα τα οποία αποτελούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τον Όλαφ και τα κρατη Μία άλλη παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή η Επιτροπή σας, μαζί με το Συμβούλιο επεξεργάζεται τον κανονισμό του Όλαφ. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν ε, συζητιέται γίνονται ακροάσεις ε, και συζητήσει με τον Επίτροπο για τον 1073 του 99 και όλα αυτά υπάρχουν στη σημείο 4 2011 της έκθεσής μας. Βασισμένη λοιπόν στην εμπειρία των τελευταίων 6 ετών έχουμε κάνει μια σειρά συστάσεων. Θα τα δείτε αυτά στην παρουσίασή μας. Πρώτα απ' όλα θα περάσω στην εποπτεία της εφαρμογής της ερευνητικής δραστηριότητας του Όλαφ. Σε όλη την περίοδο της ε, εποπτείας μας θεωρήσαμε πως αυτή η λειτουργία είναι απολύτως απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Όλαφ. Τρία σημεία θα θέλαμε να τονίσουμε. Την ε, ε, τις αρμοδιότητες του Όλαφ, την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη και την ανταλλαγή πληροφοριών με τα θεσμικά όργανα και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίε. Τα δύο πρώτα θα τα αναφέρει η κυρία Ράιτ, το τρίτο θα το κάνω εγώ. Για το πρώτο σημείο αρμοδιότητες του Όλαφ. στην ε, τοποθέτησή μας του 2010 και του 2011 εκφράσαμε πως, την άποψη πως θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ορισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του Όλαφ όπως αναφέρονται στον κανονισμό 1073 του 1999. Βεβαίως στον κανονισμό ρυθμίζεται πως έχει ο Όλαφ την, την ε, αρμοδιότητα και την ικανότητα να κάνει απροειδοποίητους ελέγχους και να έχει πρόσβαση σε όλα τα θεσμικά όργανα, στα γραφεία και στις πληροφορίες, εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι αρμοδιότητες. Δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι γνωστό και το είχαμε αναφέρει τόσο ή άλλως και το 2011. Αφορά έρευνα εις βάρος ευρωβουλευτών καθώς και πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία αμφισβητήθηκαν και τους αρνήθηκε η είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση λοιπόν την ερμηνεία του, της αρμοδιότητας του Όλαφ από ένα θεσμικό όργανο, περιορίστηκε η ανεξαρτησία του στην άσκηση των καθηκόντων του. Δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στην Κομισιόν. Ο Όλαφ μέχρι στιγμής δεν έχει άμεση και αυτόματη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των προσωπικών δεδομένων της Κομισιόν. Στην τοποθέτησή μας 1 του 2011 που συντάξαμε μετά από αίτημα του Διευθυντή του Όλαφ υποστηρίξαμε τον Όλαφ στον διάλογο αυτό με την Κομισιόν. Δεύτερον, συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη. Οπωσδήποτε η δυνατότητα επιχειρησιακής λειτουργίας του Όλαφ εξαρτάται από τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και από τη συνεισφορά τους και κατά τη διάρκεια της έρευνας αλλά και αργότερα. Όσον αφορά λοιπόν την επεξεργασία εκθέσεων για περιπτώσεις που κράτησαν πάνω από 9 μήνες είχαμε μια σειρά περιπτώσεων στις οποίες δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Επιπλέον διαπιστώνουμε τη δυσκολία που έχει ο Όλαφ να βρει τις εθνικές αρμόδιες αρχές οι οποίες θα μπορέσουν να του δώσουν την απαραίτητη βοήθεια π.χ. σε επιτόπιες έρευνες. Επιπλέον, στην σύστασή μας 4 του 2011 προτείνουμε μια αλλαγή που έχει στόχο να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να ορίσουν συνομιλητή του Όλαφ και μάλιστα ιδιαίτερα στον τομέα των άμεσων δαπανών στο επόμενο σημείο θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην συναδελφό μου την κυρία Ράιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα σχολιάσω αυτό το τελευταίο θέμα διότι δεν το κάλυψε η κυρία Τεάτο. Ε, είπε ότι για να λειτουργήσει σωστά η ΟΛΑΦ ε, χρειάζεται τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται επίσης αποτελεσματική και πλήρη συνεργασία όλων των οργανών, των φορέων, των οργανισμών της Ένωσης. Για σε πολλές υποθέσεις χρειάζεται συνεργασία όλων αυτών. Λοιπόν, η στενή συνεργασία ανάμεσα στην Όλαφε και τους εθνικούς φορείς σε βάση και των συστάσεων είναι απαραίτητο στοιχείο για να ε, ε, ευωδοθούν οι έρευνες. Ε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα λοιπόν για την ε, σωστή συνεργασία και θα πρέπει να απόσχουν όλοι από δράσεις που παρεμποδίζουν το έργο της Όλαφ. Και γι' αυτό το λόγο προβλέπεται παρακολούθηση αυτή τη διάσταση ε, των επιχειρήσεων τη Όλαφ, ε, ό,τι σχετίζεται δηλαδή με την ανεξαρτησία τη. Είδαμε ποια πρόσβαση έχει η Όλαφ πληροφορίε ε, που κατέχουν άλλοι φορεί και οργανισμοί. Συνεργαστήκαμε και με την Εσωτερική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για του Ελέγχου και άλλου οργανισμού, και εξετάσαμε και το θέμα τη παρακολούθηση των συστάσεων τη Όλαφ από πλευρά άλλων θεσμικών οργάνων. Εξετάσαμε και άλλε υποθέσει επίσης ε, όπου η Όλαφ εμποδίζει κάποιον που ε, εμπλέκεται σε μια έρευνα να γνωστοποιήσει τις ε, θέσεις του όταν ε, παραδείγματος χάρη πάγεται σε κάποιον εθνικό έλεγχο. Επίσης εξετάσαμε τη, δια... τη μέθοδο διαβίβαση των υποθέσεων από την Όλαφ και την παροχή πληροφοριών προς εθνικούς φορείς και οργανισμούς καθώς και την ανταλλαγή απόψεων με αυτού του οργανισμού. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε τέσσερι πτυχέ όλων αυτών. Πρώτον, πρόσβαση τη όλαυση τη πληροφορίε που κατέχουν άλλοι οργανισμοί και φορείς. Ε, η αποποίηση της ε, ε, του δικαιώματος του ερευνόμενου προσώπου να γνωστοποιήσει τις απόψεις του πριν το πέρας της έρευνας, διαβίβαση των υποθέσεων από πλευράς της Όλαφ. Θέλω να περάσω στο πρώτο θέμα σε σχέση με την, παροχή των πληροφορι... την πρόσβαση των πληροφοριών από πλευράς της Όλαφ υπάρχουν κάποιες υπόνοιες υποψίες ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με την πρόσβαση της Όλαφ σε βάσεις δεδομένων που κατέχουν άλλα θεσμικά όργανα όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο άρθρο 4, εδάφιο 2 του κανονισμού 1073 στο πρώτο τμήμα αναγνωρίζεται σαφώς το δικαίωμα της ε, Όλαφ χωρίς πρώτερη ειδοποίηση να κατέχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ε, που έχουν άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φάνη ιδιαίτερη απρόθυμη να δώσει τα και ε, ε, απρόσκοπτη πρόσβαση σε διάφορε βάσει δεδομένων και αρχεία και έτσι παραβιάζεται ο κανονισμό 45 ε, του 2001, δηλαδή ο κανονισμό περί προστασία των δεδομένων. Χρειάζεται πρόσβαση όλα σε τέτοιου είδου πληροφορίε, κυρίω στι αρχικέ φάσει τη έρευνα, προτού συνταχθεί Φάκελο ε, Έρευνα, για να αποφασίσει ποια θα είναι και τα κριτήρια που θα εφαρμόσει στην έρευνα που κάνει. Ε, και έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση. Βάσει τις συστάσεις που κάναμε το 2011 και χάρη στον ε, προϊόν διάλογο ανάμεσα στην Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζουμε πια ότι ε, στο εγγύς μέλλον θα έχουμε κάποια λύση. Ο τροποποιημένος κανονισμός επίσης θα καλύψει αυτά τα θέματα, επιτυγχάνοντας μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη της Όλαφ να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες όλων των θεσμικών οργάνων πριν να ανοίξει έρευνα και στα ε, πρωταρχικά στάδια αυτή. Ε, ισορροπή λοιπόν ανάμεσα σε αυτό και την κείμενη νομοθεσία περί προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, όταν κάποιο αποτελεί αντικείμενο έρευνα, παρεμποδίζεται από την Όλαφ ε, να γνωστοποιήσει τι θέσει του. Όταν διεξάγεται η έρευνα, χρειάζεται πρώτερη συγκατέθεση από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Φορέα του θεσμικού οργάνου για να παρακάμψει αυτόν τον κανόνα και να ε, ε, επιτρέψει στον ε, υποέρευνα άνθρωπο να γνωστοποιήσει τις απόψεις του. Το 2010 στις συστάσεις μας είπαμε ότι όταν παρακολεί ή παρεμποδίσει τη διαδικασία ένα θεσμικό όργανο τότε τίθεται σε κίνδυνο το έργο της Όλαφ και τα αποτελέσματα του ελέγχου και σε πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι παρεμποδίστηκε η διαβίβαση αυτών των υποθέσεων στη, στους εθνικούς φορείς λόγω της καθυστέρησης που αποδίδεται σε αυτούς τους φορείς. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτον, ο Γενικός Γραμματέας ενός οργάνου καθυστέρησε 14 μήνες μέχρι να δώσει την έγκρισή του στο αίτημα της ε, Όλαφ παρότι <clears throat> παρά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα, χωρί καν κάποια αιτιολόγηση. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εν λόγω Γενικό Γραμματέα, ε, μετά από αρχική απόρριψη του αιτήματο, ε, εκχώρησε την έγκρισή του, όμω μετά από την πάροδο πέντε μηνών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό ε, κίνδυνο παρακόλληση προϊόντων ερευνών λόγω ε, της ε, ε, άρνηση του αιτήματο να επιτρέψει η Όλαφ στο έρευνα άτομο να γνωστοποιήσει τις απόψεις του. Λοιπόν, ο νέος τροποποιημένος κανονισμός έχει τις κατάλληλες διατάξεις για να αποφύγουμε τέτοιου είδους περιστατικά στο μέλλον. Ε, και ο τρόπος με τον οποίο ε, έχει, ε, ρυθμίζεται ε, αυτό το θέμα στον τρέχοντα κανονισμό, το 1043 δεν είναι ικανοποιητικός. Τρίτον, η υποχρέωση από πλευράς της Όλαφ να χορηγεί πληροφορίες στα διάφορα όργανα και οργανισμούς. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας έχει νομική υποχρέωση η Όλαφ να ενημερώνει τα θεσμικά όργανα σε περίπτωση που ο εσωτερικός ελεγχός καταδεικνύει ότι μπορεί να εμπλέκεται και ένα μέλος του μόνιμου προσωπικού. Υπάρχει βέβαια και εξαίρεση όταν υπάρχει υποχρέωση απόλυτη εμπιστευτικότητα για του στόχου τη έρευνα ή διότι οι έρευνε υπάγονται στην αρμοδιότητα μια εθνική δικαιοδοτική αρχή. Το άρθρο 4.6 του τροποποιημένου κανονισμού ε, τροποποιεί αυτού του κανόνε και αναφέρει ότι σε έκτακτε περιστάσει, ε, όταν η εμπιστευτικότητα τη έρευνα δεν μπορεί να κατοχυρωθεί με διαφορετικό τρόπο, η Όλαφ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ε, πρόσφορε εναλλακτικέ οδού για να προμηθευτεί τι πληροφορίε. Πριν το 2011 Είχαμε εκφράσει ανησυχία μας για αυτό το θέμα και θεωρήσαμε ότι ε, λόγω αυτής της διάταξης ε, τη τη διακριτική ευχέρεια της ε, Όλαφ να διατηρούν την εμπιστευτικότητα όταν όμως κρίνουν οι εκπρόσωποι της Όλαφ ότι είναι αυτό απαραίτητο. Τέταρτον, ε, ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι η διαβίβαση των τελικών ε, φακέλων σε εθνικούς φορείς, οργανισμούς ή θεσμικά όργανα. Η Όλαφ αποφάσισε να κατόπιν αιτήματο Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στείλει όλες, ε, όλους τους φακέλους προέκυψαν από εσωτερικούς ελέγχους ε, στα πλαίσια αυτής της ε, παρακολούθησης. Επιπροσθέτως αποφάσισαν να εφαρμόσουν την ίδια πολιτική και για λοιπούς οργανισμούς και όργανα εκτός αν υπάρχει αντίθετο αίτημα. Λοιπόν, εξετάζαμε αυτή την πρακτική για να διαπιστώσουμε αν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Όλαφ κατά την επιτέλεση του ερευνητικού του έργου και στην σύσταση 5 του 2011 εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι αυτή η διαβίβαση των φακελών μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα των εμπλεκομένων σε αυτή την έρευνα και μπορεί να οδηγήσει ε, σε αγωγέ για αποζημίωση ενώπιον του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ε, θα πλήξει την αξιοπιστία και τη φήμη και το κύριο ε, τη Όλαφ. Η διαβίβαση των φακέλων με ευαίσθητε πληροφορίε σχετικά με μάρτυρε, πληροφοριοδότε κτλ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την έκβαση της ε, ε, έρευνας ε, γιατί δεν επιτρέπει στην Όλαφ να επιτελέσει την έρευνα. Δεχόμαστε 100% τις παρατηρήσεις ε, που έγιναν ε, μετά από την έκδοση αυτής της νομοδότησης από τον ε, ίδιο τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον εκπρόσωπο της Όλαφ. Βάσει αυτών των συστάσεων όλοι οι φάκελοι, είτε υπάρξει παρακολούθηση ή όχι, θα πρέπει να διαβιβάζονται, συμφώνησαν όλοι, όμως αυτό δεν συμβαίνει ότι όλα τα στοιχεία του τελικού φακέλου πρέπει να διαβαστούν, ε, μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να προσαρμόσουμε την έκθεση και να αφαιρέσουμε τα ευαίσθητα ε, στοιχεία σε περιπτώσεις βεβαίως όμως που εμείς εξετάσαμε. Δεν έγινε αυτό. Αυτή η πρακτική νομίζω θα προσφέρει ε, μέσα σε άλλους θεσμού για την παρεμπόδιση του ερευνητικού όργου της Όλαφ, υπονομεύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού προς την αξιοπιστία και το κέρδος τη Όλαφ. Άρα προτείνουμε να αναθεωρήσει η Όλαφ την απόφασή για την διαβίβαση ε, των εκθέσεων όπως είναι χωρί ε, χωρίς επεξεργασία στους ε, μπλεκόμενους φορείς. Θα πρέπει να αναλυφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε η πρακτική που ακολουθείται να συνάδει με την ε, νομοθεσία της Ένωσης και να μην θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχοντες. Θα ήθελα να περάσω τώρα ε, στα, στις επιπτώσεις ε, του, της διαχείρισης αυτών των ερευνητικών αρμοδιοτήτων ε, της Όλαφ πιστεύουμε ότι αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να υπάγονται σε πλήρη ανεξαρτησία ως προς τη διαχείριση των ερευνών, ως προς τον προγραμματισμό, το στρατηγικό προσανατολισμό αυτών, τον μηχανισμό, ε, ούτως ώστε ε, να ελέγχεται εσωτερικά η δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια της και φυσικά έλεγχος της νομιμότητας ε, των δραστηριοτήτων. Εδώ εμπλέκονται και θέματα καταστατικού προσωπικού, διότι μιλάμε για ερευνητικές αρμοδιότητες της Όλαφ ε, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι υπάρχει ένα σχετικό εγχειρίδιο πλέον στην Όλαφ ε, σε διάφορες νομοδοτήσεις που έχουμε εκδώσει σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού ε, η Οπτική Επιτροπή τόνισε επανειλημμένα ότι το βασικό μέτρο που πρέπει να αναλάβουμε για να κατοχυρώσουμε την ανεξαρτησία της Όλαφ της έρευνας ε, είναι η χορήγηση επαρκών κονδυλίων στην Όλαφ. Επαρκή κονδύλια πρέπει να εξασφαλίζονται πάντοτε φυσικά σε περίοδους οικονομικής ύφασης χρειάζονται δημοσιονομικοί περιορισμοί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Όλαφ δεν είναι στο απειρόβλητο βέβαια, ε, αλλά ένα ανεξαρτικό, ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο χρειάζεται να είναι ανεξάρτητο επίση και από πλευρά προπολογισμού. Βάζει τη σύσταση 3 του 2011 ο Γενικό Διευθυντή τη Όλαφ και μόνο πρέπει να έχει την δυνατότητα να αποφασίσει οι ενδεχόμενε περικοπέ του προπολογισμού βάσει το οποίο λειτουργεί η Όλαφ. Now pass Να περάσω τώρα στις νομοθετικές διατάξεις περί εγγύησης της ανεξαρτησίας του Όλαφ. Όπως ξέρετε υπάρχουν δύο εγγυήσεις για την εγγύηση της ανεξαρτησίας του Όλαφ. Πρώτον, την ανεξαρτησία του Γενικού Διευθυντού και δεύτερον, την ανεξαρτησία της Εποπτικής Επιτροπής. Η ανεξαρτησία του Γενικού Διευθυντού είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση γιατί έτσι δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα επιρροή στις διοικητικές έρευνες. Σε μια σειρά τοποθετήσεων η Εποπτική Επιτροπή εξέφρασε την άποψή της για τον ορισμό του Γενικού Διευθυντού, για τις δυνατότητες να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του και για το ζήτημα της αναπλήρωσής του. Θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο τελευταία σημεία την διασφάλιση δηλαδή της ανεξαρτησίας. Υπενθυμίζω πως μόνο ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να αποφασίσει για την έναρξη και διεξαγωγή ερευνών χωρίς εξωτερικές οδηγίες από κανέναν. Η δυνατότητα καταγγελίας κατά της Κομισιόν όταν υπάρχει ε, κάποια τέτοια παραγγελία μπορεί να αμφισβητήσει την εξαρτησία του Όλαφ. Με βάση λοιπόν τις τελευταίες αυτές νομοθετικές διατάξεις στη σύστασή μας υπαριθμών 4 του 2011 προτείνουμε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβαση και έρευνα σε όλα τα θεσμικά όργανα και αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις κομισιών μπορεί να λειτουργήσει ως αρχή προσλήψεων ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ. Εμείς θεωρούμε πως το ερευνητικό προσωπικό του Όλαφ μπορεί να τοποθετηθεί από τον Διευθυντή χωρίς να ακολουθηθεί η μακροσκελής διαδικασία που ακολουθείται για το λοιπό προσωπικό της Κομισιόν. Το ζήτημα του αναπληρωτή Διευθυντού επίσης μας απασχόλησε. Σύμφωνα με την πρώτο Γενικό Διευθυντή της ε, Όλαφ, η Κομισιόν είχε ορίσει κάποιον προσωρινό ε, γενικό διευθυντή, αλλά εμείς θεωρούσαμε πως θα έπρεπε να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή για να υπάρχει μια συνέχεια στην διοίκηση. Όσον αφορά τώρα τον ρόλο της Εποπτικής Επιτροπής, θα ήθελα να πω πως η ανεξαρτησία της Εποπτικής Επιτροπής είναι σημείο κλειδί για την επιχειρησιακή ανεξαρτησία του Όλαφ. Για να μπορέσει η Επιτροπή αυτή να επιτελέσει τον ρόλο της θα πρέπει τα μέλη της να είναι επαρκή όπως ανέφερε και κατερτισμένα όπως ανέφερε και η συναλφός μου. Το ίδιο ισχύει και για την γραμματεία που διατίθεται από τον Όλαφ η οποία θα πρέπει επίσης να έχει ικανό αριθμό αλλά και να είναι στελεχωμένη από άτομα με τις ανάλογες δεξιότητες. Δυστυχώς το νέο οργανόγραμμα, όπως ξέρει και ο κύριος Κέσλερ, προβλέπει μείωση των θέσεων. Η Εποπτική Επιτροπή καταλήγει στην εκτίμηση πως προσεχώς το προσωπικό της γραμματείας αυτής θα μπορούσε να προέρχεται από άλλες υπηρεσίες πλην όλα. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει η ανεξαρτησία της Επιτροπής Εποπτείας και της Γραμματείας αυτής και αυτό κατά την απόψή μας σημαίνει πως δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τον οργανισμό τον οποίο θα πρέπει να επιβλέπει. Συμπεράσματα σύντομα στην... στις εκθέσεις μας μέχρι τώρα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή για την ανεξαρτησία του Όλαφ. Στην τελευταία αυτή έκθεση δραστηριότητας διαπιστώνουμε όμως μια σειρά κινδύνων και επηρεασμών της, δραστηριο... της ανεξαρτησίας αυτής. Δεν φτάνουμε στο σημείο να λέμε πως υπάρχει κάποια πρόθεση να ε, βλαφτεί η ανεξαρτησία του Όλοφ. Τα, παράδειγμα, τα παραδείγματα αυτά, με συγχωρείτε όμως, που αναφέραμε ε, δείχνουν πως μπορεί να υπονομευθεί αυτή η ανεξαρτησία στην πράξη. Τέλος, το συμπέρασμά μας είναι πως η ανεξάρτητη λειτουργία του Όλαφ μπορεί να διασφαλιστεί όταν διασφαλίζεται και η ανεξαρτησία της Εποπτικής Επιτροπής. Η κυρία Ράιτ και εγώ προσπαθήσαμε στον ρόλο μας αυτό να είμαστε επικριτικοί φίλοι του Όλαφ και σας ευχαριστούμε για την προσοχή μας και να προσθέσω κύριε Πρόεδρε, σας συγχαίρω για την ε, εκλογή σας στην Προεδρία της Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ja, vielen Dank, Frau Wright, und vielen Dank, Frau Ευχαριστώ κυρία Ράιτ, κυρία Τεάτο για την έκθεση, για το έργο σας και με τη λήξη της θητείας σας νομίζω μπορούμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Εσάς και ολόκληρη την Εποπτική Επιτροπή. Συμφωνήσαμε τώρα πως θα ακούσουμε έναν γύρο ερωτήσεων Θα δώσω πρώτα απ' όλα λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια Ingeborg Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Εποπτική Επιτροπή και τις δύο κυρίες που ήρθαν σήμερα το πρωί. Αυτά τα οποία είπαν ήταν ήδη ανησυχητικά για την Επιτροπή μας, η οποία βεβαίως θεωρούμε πως είναι ακριβώς ο προστάτης Άγιος της καταπολέμησης της απάτης. Βλέπουμε λοιπόν το φαινόμενο αυτό το οποίο εμφανίζεται και το θέμα αυτό της νομικής βάσης το έχω θίξει πάρα πολλές φορές στον τριμερή διάλογο και ε, από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να υπολογίζουμε σε ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να υποστηρίξω λοιπόν την Εποπτική Επιτροπή στη διαπίστωσή της για κινδύνους επηρεασμού αλλά και της σταδιακής υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του Όλεφ. Τα είπε νομίζω αρκετά επαρκώς η Επιτροπή, οπότε εγώ θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε κάποια σημεία στα οποία θεωρώ πως εμείς ως αρχή προϋπολογισμού και ως νομοθέτης ε, πρέπει να έχουμε λόγο. Ας ξεκινήσουμε με την ίδια την Εποπτική Επιτροπή. Η Εποπτική Επιτροπή είχε μείωση του προσωπικού, έχει αυτή τη στιγμή πέντε διοικητικά στελέχη και τρία στελέχη γραμματείας. Είχαν πει οι άνθρωποι, έχουν 8 άτομα, είχαν πει δε, πριν από λίγα χρόνια ότι ήθελαν 10 Ήδη δηλαδή το ότι είχαν περιοριστεί στα 8 ήταν θυσία. Τώρα να περιοριστούν κι άλλο στη γραμματεία τους είναι πάρα πολύ. Δεν το θεωρώ σωστό αυτό γιατί ο Όλαφ ε, ούτως ή άλλως πέρσι είχε 5 εκατομμύρια αδιάστα κονδύλια τα οποία επέστρεψε στην Κομισιόν. 5 ε, εκατομμύρια νομίζω ε, στα 40 εκατομμύρια διοικητικό κόστος είναι πάνω από 10 100. Ε, Τώρα, εάν μιλήσουμε για πρόσληψη προσωπικού πρέπει να υπενθυμίσω τον κανονισμό της ίδιας της Επιτροπής Εποπτείας που μπορείτε να τον διαβάσετε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου αναφέρεται πως έχει λόγο η Επιτροπή στην στελέχωσή της. Και αυτό το δικαίωμα συναπόφασης δεν δόθηκε ποτέ στην Επιτροπή. Ε, δεν γίνεται αγαπητοί φίλοι. Τι κάνουμε δηλαδή. Λυπούμε, δεν, δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς θα γίνουν τα πράγματα στο μέλλον. Κατόπιν να έρθω σε αυτό το οποίο θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει, δηλαδή το θέμα του πώς εργάζεται η υπηρεσία. Η Εποπτική Επιτροπή διαπιστώνει στην έκθεσή της πως έχουμε το πρόβλημα της παραγραφής και της μη ε, εμπλοκής ε, εθνικών εμπρογνωμών. Στον κανονισμό 9 παράγραφος 2 αναφέρεται σαφώς πως θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εθνική νομοθεσία ε, ο Όλαφ. Δηλαδή, τι νόημα έχει να συγκεντρώνει στοιχεία που δεν μπορεί μετρά να παρουσιάσει στο δικαστήριο. Αυτό είναι βασικό και έχει για εμάς ως ε, κοινοβούλιο ε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μην ξεχνάτε, μου είχαν δείξει εμένα στατιστικά στοιχεία του 2009 πως 93% ε, των ερευνών του Όλαφ καταλήγουν στον γκάδο ανακύκλωσης γιατί, γιατί δεν μπορεί να δοθεί καμία συνέχεια. Οπότε, αν δεν συμβαίνει τίποτα τελικά, ή έχουμε πρόβλημα. Είπαμε πως θα κάναμε έναν έλεγχο νόμιμότητας που θα έπρεπε να μπει αυτομάτως στη λειτουργία του Όλεφ. Αυτό το έχουμε γράψει μόνο μέχρι στιγμής στον κανονισμό στις ε, τροπολογίες. Βλέπουμε τώρα στο νέο οργανόγραμμα πως από το Φεβρουάριο του 2012 οι θέσεις οι οποίες είχαν προβλεφθεί γι' αυτό διαγράφονται. Και λέγεται πως αντικαθίσταται από έναν ε, έλεγχο αρχικό. Ε, δεν μπορεί νομίζω να το αντικαταστήσει αυτό εξακολουθεί να παραμείνει ανοιχτό και άλλο αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στις δύο κυρίες στην Εποπτική Επιτροπή πώς το κρίνουν, τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα, ειδικά και σε σχέση με την τελευταία οργανωτική μεταρρύθμιση. Κάτι πρέπει να γίνει κατόπιν. Να ευχαριστήσω την Εποπτική Επιτροπή για τις διαπιστώσεις της για αυτή την σταδιακή μείωση των δικαιωμάτων του Όλαφ και των διοικητικών ε, προσκομμάτων ε, που αντιμετωπίζει. Το ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, είναι ευαίσθητα βεβαίως για τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων τους, εντάξει, είναι λογικό. Αλλά το εάν επιτρέπεται το αποτέλεσμα μιας έρευνας να πάει στις εθνικές αρχές ή όχι, όχι δεν είναι δυνατόν. Δεν ρωτάει κανένας ε, έναν απλό πολίτη του ε, κράτους μέλους ή έναν υπάλληλο του κράτους μέλους το εάν θα πάει η υπόθεσή του στην δικαιοσύνη, αλλά εδώ πέρα ρωτάνε τον υπάλληλο το εάν ε, ε, το εάν συμφωνεί ο επικεφαλής, μάλλον δεν τον τον επικεφαλής της υπηρεσίας του, το, εάν θα πάει η υπόθεση αυτή στι αρμόδιες αρχέ. ή όχι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση και όχι να αποφασίζουμε κατά περίπτωση, γιατί και εδώ πέρα πρέπει να το δούμε αυτό στη μεταρρύθμιση του Όλαφ. Το είπαμε, θέλουμε ίση μεταχείριση για όλου αλλιώ δεν γίνεται. Ε, και εδώ πέρα συμφωνούμε πλήρως. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε κάτι τέτοιο, να έχουμε διαδικασίες οι οποίες καθυστερούν επί 15 μέρες γιατί αρνείται, δεν, αρνείται ένα θεσμικό όργανο να δώσει τα αποτελέσματα της έρευνας στις εθνικές αρχές. Και μετά επέρχεται η παραγραφή κτλ. Εδώ πέρα νομίζω σωστά το κάναμε και ξεκαθάρισαμε το τι θέλουμε. Τώρα, πρόσβαση στις τράπεζες δεδομένων της Κομισιόν. Ναι, πράγματι σημαντικό. Θέλουμε να υπάρχει η εγγύηση, α, η πρόσβαση άμεση, εγγυημένη και αυτόματη. Ε, βεβαίως υπάρχει και ο επόπτης προσωπικών δεδομένων, στον οποίο υποβάλαμε μια σχετική διατύπωση ακόμα βεβαίως δεν πρόλαβα γιατί είχα και ζήτημα με κάποια άλλη δουλειά που κάνω παράλληλα, αλλά νομίζω πως αυτό το ζήτημα πρέπει και μπορεί να λυθεί, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε καθόλου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του Όλαφ. Για τη γνωμοδότηση τώρα υπαριθμών 5 του 2011. και εκεί πέρα συμφωνούμε πλήρως με την Εποπτική Επιτροπή για τα εμπόδια που υπάρχουν σε κάποιον, σε κάποιον καταγγέλλοντα. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει και εδώ πέρα να βρεθεί μια λύση. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη επίθεση που υπάρχει στις καταγγελίες μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να βασιστεί σε κάποια εμπιστευτικότητα ο καταγγέλων. Ε, πρέπει να γίνει κάτι κατεπηγόντως εδώ πέρα να αναφερθώ επίσης στο τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος με τον κανονισμό. Πρέπει να λύσουμε κάποια ε, ζητήματα ε, για τη συνέχεια των εργασιών. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής είναι δύσκολο ζήτημα και νομικά πρέπει να βρεθεί ε, μια λύση. Αυτό το οποίο προτείνει η Εποπτική Επιτροπή, δηλαδή δικαίωμα καταγγελίας κατά όλων των θεσμικών οργάνων, ναι, συμφωνούμε απολύτως. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε, υπάρχουν κάποια θεσμικά προβλήματα, γιατί ο Όλαφ ε, είναι τμήμα της Κομισιόν και το θέμα μετά ποιος εκπροσωπεί την Κομισιόν σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχει ακόμα λυθεί. Τώρα, για έρευνε κατά βουλευτών. Εδώ πέρα διαφωνώ με την Εποπτική Επιτροπή. Γιατί ο κανονισμός του Όλαφ νομίζω δεν μπορεί να παραβιάσει το πρωτογενές δίκαιο. Και το πρωτογενές δίκαιο λέει πω υπάρχει βουλευτική ασυλία. Βλέπουμε βεβαίω με μεγάλη ανησυχία πως τα τελευταία δέκα χρόνια δεν γίνεται σεβαστή η βουλευτική ασυλία και με τις τωρινές διαδικασίες. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά, απλά το λέω. Δηλαδή, όταν έχουμε ασυλία, πρέπει να λαμβάνεται και υπόψη αυτή. Είναι ένα αγαθό το οποίο, ε, ένα προνόμιο το οποίο έχει εγγραφεί στις συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν να, να παραβιάσουμε τις συνθήκες και να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που γράφουν. Ε, και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει για να μην χρειάζεται να έχουμε διαφωνίες στο μέλλον. Να διαβεβαιώσω δε την Εποπτική Επιτροπή πως εκτιμούμε το έργο της και την εμπειρία της, γιατί γίνεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή όπου έχουμε το νέο κανονισμό, τη συζήτηση για το νέο κανονισμό και χρειαζόμαστε την εμπειρία της Επιτροπής. Γι' αυτό ελπίζω εποπτική επιτροπή του Όλαφ με τη νέα της σύνθεση να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί το στομότερο δυνατόν. Και να υπενθυμίσω και την νέα εποπτική επιτροπή πως είμαστε φίλοι σε αυτή την επιτροπή γιατί ούτως ή άλλως λειτουργεί δύο οργανικά υποπτική επιτροπή και ούτως ή άλλως ε, πρέπει να συνεργαζόμαστε ακριβώς γιατί πρόκειται για τον εγγυητή της ανεξαρτησίας του όλαφου, ο οποίος προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι στις δύο συναδέλφους καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στο μέλλον. Θεωρώ πως ε, επιτελέσατε πάρα πολύ καλά το έργο σας και συνεισφέρατε στο κύριο της ε, Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε περνάμε τώρα στην συζήτηση. Ο κύριος Μπαλτσίτης έχει πρώτο το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ε, σας ευχαριστήσω για την ε, λεπτομεριακή παρουσίαση ενός πολυσχηδούς θέματος στην Επιτροπή και θα ήθελα Επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Ίγκεμπορ Γκρέσλε, την εισηγήτρια, για την παρουσίαση αυτή, την λεπτομεριακή αυτή παρουσίαση. γιατί μας παρουσίασε λεπτομερώς την εκθέση αυτή. Στα πλαίσια των ε, σκιωδών θα ήθελα να πω ότι ε, λυπούμεθα γιατί δεν μπορέσαμε να συμμετάσχουμε σε όλη τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και των ε, διεργασιών. Εγώ συμμετέχω σε αυτή την επιτροπή για περισσότερα από δύο χρόνια και αντιμετωπίσαμε ε, και εξετάσαμε πολλές εκθέσεις. Η μία υποβλήθηκε από την Κομισιόν. Στη συνέχεια συζητήσαμε τις εκθέσεις της Όλαφ και έχουμε μία επανάληψη των δεδομένων. Μιλάμε για την ανεξαρτησία της Όλαφ και αυτό είναι το ε, σημαντικό μας θέμα. Θέλουμε και λεπτομέρειες από όλα τα κράτη. Όταν ε, η Επιτροπή ε, δημοσιεύει την έκθεσή της, αναφέρεται στο γεγονός ότι όλα τα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα, διότι τα κράτη-μέλη δεν μας ε, παραχωρούν όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος, ο οποίος όλο ένα και συνεχίζεται. Η Όλαφ ποτέ δεν θα είναι ανεξάρτητη παρά μόνον όταν φτάσουμε σε ένα ανεξάρτητο σύστημα πρόσβασης δεδομένων. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ιστορία και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να είναι ιδιαίτερα δραστήρια και να μας πει ποιες είναι οι προαπαιτήσεις για την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική νομική δομή και δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προαπαιτήσεις ε, πάντα. Και ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν καν να δώσουν τα στοιχεία αυτά στην Κομισιόν. Θα πρέπει επίσης να αλλάξει το θέμα της ευθύνης και της λογοδοσίας. ο κύριος Σεμέτα θα πρέπει να ανησυχήσει κάπως, διότι τη στιγμή που η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή δεδομένων από όλα τα κράτη-μέλη, ε, σύντομα 28, τότε θα παραμένουμε στο ίδιο θέμα, στο αρχικό τετραγωνίδι, ότι δηλαδή τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να τα δεν είναι συγκρίσιμα, γιατί οι εξειδικευμένοι οργανισμοί στα κράτη-μέλη διαφέρουν. Στη Λιθουανία υπάρχουν πέντε τέτοιοι οργανισμοί, δεν ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους και βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτή τη μικρή χώρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι κατά πόσο η Κομισιόν δεν θα πρέπει να ορίσει ένα σύστημα ή να αλλάξει τις ε, νομικές απαιτήσεις. Γιατί όταν προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αλλάξαμε άρδιν και το νομικό μας ε, πλαίσιο, τη νομική πλαισίωση. Αυτό αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την ίσπραξη φόρων, αλλά δεν μιλήσαμε για την προστασία των χρηματοοικονομικών μας ε, συμφερόντων, διότι το οργανωμένο έγκλημα προσπαθεί να εξεύρει τρόπους έτσι ώστε να υποκλέπτει ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε και προαναφέρθηκε το 1994, μας απασχολεί από τότε και γι' αυτό θα πρέπει να αναλυθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει βεβαίως ένταση μεταξύ της Εποπτικής Επιτροπής και της ΟΛΑΦ άλλαξε ο Γενικός Διευθυντής, γίνεται μία μεταρρύθμιση του οργανογράμματος και της οργάνωσης και πολλά στοιχεία θα πρέπει να, να αλλάξουν εμείς ως μέλη αυτής της Επιτροπής. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες στο μέλλον για να έχει η όλα αυτή κατάλληλη χρηματοδότηση, γιατί χωρίς χρήματα δεν μπορεί να φτάσει και σε αυτά αποτελέσματα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Όλαφ θα πρέπει αρχικά να εστιάσει την προσοχή της στις έρευνες οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι τόσο χρονοβόρες και να είναι πιο αποδοτικές και βεβαίως απότερο στόχος είναι να φτάσουμε στα απαραίτητα στοιχεία. Εν κατακλείδη θεωρώ ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο για την ε, εποπτική αρχή και θα πρέπει να προστατεύσουμε τα χρηματοοικονομικά μας συμφέροντα. Με κοινέ προσπάθειες θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πιο κεντρικό σύστημα το οποίο θα ε, ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Και όσο το νωρίτερο, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία παντού. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για χρηματοοικονομικές απάτες ή παρατυπίες. Θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές σύστημα πρόσβασης στα δεδομένα και λογοδοσίας. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Der nächste ist der äh, Kollege Paul Rübig, bitte. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Ναι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχει την απαραίτητη πρόσβαση και η Υποπτική Επιτροπή. Ξέρουμε βεβαίως με την κυρία Τεάτο πως έχουμε καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο πάντα και ούτως ή άλλως το Κοινοβούλιο δημιούργησε τις συνθήκες ύπαρξης του Θυμάμαι πως είχαμε παλέψει ο Όλαφ να έχει μια σωστή νομική βάση. Και βεβαίως η εποπτεία μιας τέτοιας αρχής ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη και κεντρική σημασία και ειδικά σε καιρούς ε, κρίσης και κρίσης χρέους είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την διαφάνεια της λειτουργίας. Για μένα τώρα είναι σαφές, πρέπει να αναφερθούμε νομίζω και στην σύγκρουση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πως οι βουλευτές έχουν ε, ασυλία και δεν είναι ε, για πλάκα αυτό το πράγμα. Ο βουλευτής εκπροσωπεί ένα τμήμα του ε, πληθυσμού, του λαού ούτως ή άλλως. Και ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει πάρα πολλά πράγματα στην ε, δραστηριότητά του ως πολιτικός ε, χρειάζεται αυτή την ασυλία και εδώ πέρα συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε πως ειδικά ε, σε καιρούς προεκλογικούς δεν πρέπει να δίνουμε εφόδια στους ανθυποψηφίους ενός βουλευτή. Γιατί ξέρετε πως όταν συμβαίνει κάτι στο κοινοβούλιο αμέσως τρέχουν, ενώ κάτι δυσάρεστο, τρέχουν τα ΜΜΕ γιατί ε, δημιουργεί θόρυβο και βεβαίως μετά από δύο χρόνια κανένας δεν μαθαίνει το ότι ήταν αθώος ο βουλευτής, η ζημιά έχει γίνει και είναι ανεπανόρθωτη. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει ε, και η Εποπτική Επιτροπή να έχει επαφές με τα κράτη-μέλη. Τι κάνετε ως προς αυτό, υπάρχουν πληροφορίες ε, ή απλά επικεντρώνεστε στη βασική λειτουργία του Όλαφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυλακάκης έχει το λόγο. Thank you, uh, Mr. President and, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εύχομαι να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές σας. Αν κοιτάξει κανείς ε, σε τι πρέπει να μας βοηθά ιδανικά η Εποπτική Επιτροπή, διαπιστώνει ότι ορισμένε φορέ πρέπει να περιοριζόμαστε στα βασικά. Ποια είναι τα βασικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλούστατα. Ε, πόσες απάτες, ε, σε ποιο ποσοστό οι απάτες αυτές υπάρχουν στην αρμοδιότητα της Όλαφ. Έχουμε κάποια εικόνα γι' αυτό, δεν νομίζω. Ε, πόσες απάτες ε, εκθέτουμε. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Πολύ λίγα. Αυτά είναι βασικά δεδομένα ε, στη συζήτηση που κάνουμε. Με πόση αποτελεσματικότητα τώρα διαχειριζόμαστε τους σπόρους της Όλαφ. Εγώ προσωπικά πιστεύω όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, αλλά όχι λόγω του, της μεθοδολογίας εργασίας της Όλαφ. Σε πολλές περιπτώσεις και εξάλλου αυτό μας λέει η Εποπτική Επιτροπή, αυτό οφείλεται στα σοβαρά κολλήματα που προέρχονται όμως από όλους τους υπολείπους πέραν της Όλαφ. Αδυναμία πρόσβαση στις πληροφορίες, κάποιοι προσπαθούν να παρακολύσουν τις έρευνες, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δηλώσουμε ευχαριστημένοι με τα τωρινά αποτελέσματα. Αυτή είναι και η πρώτη μου παρατήρηση. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και με ποιο τρόπο η Εποπτική Επιτροπή η επερχόμενη μπορεί να μας επικουρήσει. Πρώτον, ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σχηματίσουμε μία εικόνα για την έκταση της ε, απάτης, ε, της περιπτώσεις ε, όπου διαπιστώνεται απάτη. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό για να αποφασίσουμε αν η Όλαφ κάνει καλά ή όχι την δουλειά της. Δεύτερον, θα πρέπει να δώσουμε και τα πετούμενα μέσα στην Όλαφ για να κάνει την δουλειά της και έρχομαι απευθείας στα κονδύλια που δίνουμε στην Όλαφ. Όταν άκουσα τη συνάδελφο Γκρέ Πρέσλε να λέει ότι επιστρέφονται από την Όλαφ κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, χτύπησε ένα καμπανάκι μέσα μου. Τι σημαίνει αυτό, δεν τα χρειάζεται ή δεν έχει τρόπο να τα διαθέσει. Εγώ θα περίμενα, θα υποψιαζόμουν ότι θα ζητούσε περισσότερα κονδύλια η Όλαφ για να έχει ακόμη περισσότερα αποτελέσματα. Ε, ε, χάρη σε αυτά τα νέα κονδύλια και πολύ θα χαιρόμουν αν αυτό συνέβαινε. Θα ήθελα τώρα να περάσω κάποια ειδικότερα θέματα. Ασυλία. Πιστεύω πως ε, δεν θα πρέπει ε, να τέθεται να αμφιβόλω ούτε η ασυλία αλλά ούτε και η διαφάνεια. Άρα θα πρέπει ε, οι αρχές εδώ του Κοινοβουλίου να συνεργαστούν με την Όλαφ με τρόπο ώστε να μην αμφισβητείται η αρχή της ασυλίας αλλά και να μην παρεμποδίζονται οι έρευνες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Δεύτερον, η πρόσβαση της Όλαφ σε έγγραφα ανθρώπους που πρέπει να ε, ανακρίνει κτλ. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο, χωρίς καμία αιτιολόγηση, να υπάρχουν τέτοια κολλήματα, δηλαδή πέρα από το λόγο ότι κάποιοι δεν θέλουν να μπει στα χωράφια τους ή όλα. Μα δεν είναι δικά τους τα χωράφια, είναι των πολιτών της Ένωσης. Ε, Τρίτον, όσοι καταδίδουν, όσοι ε, καταγγέλουν, συγγνώμη. Ε, ο τρόπος ε, που χειριζόμαστε ε, αυτούς τους ανθρώπους οδηγεί σε μείωση του αριθμού τους. Άρα θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να προστατεύσουμε καλύτερα όσους καταγγέλνουν τα κακώς ε, ε, κείμενα. Τέλος, ένα άλλο ζήτημα που έχει σημασία κατά τη γνώμη μου, ποιο ποσοστό των ερευνών της Όλαφ ξεκινούν βάσει κάποιας καταγγελίας και ποιο ποσοστό ε, γίνεται αυτεπαγγέλτος ε, βάσει πρωτοβουλίας της Όλαφ. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε αν βεβαίως έχετε τα σχετικά στοιχεία μαζί σας ή μπορεί να έχετε ήδη διαμορφώσει άποψη γι' αυτό. Ε, το ερωτώ διότι οι έρευνες που βασίζονται σε πρωτοβουλία της Όλαφ έχουν ιδιαίτερη σημασία για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά της. Ε, δηλαδή, αυτός που καταγγέλει τα κακό κείμενα, ε, τα καταγγέλει γιατί κάτι πήγε στραβά. Το, η οργανωμένη εγκληματικότητα δεν έχει λοιπόν τέτοιους ε, ανθρώπους, ε, δεν υπήρχε κάποια διαδικασία που δεν λειτουργήσε αισίως και ούτως ή άλλως ε, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί ο αριθμός ε, αυτών που καταγγέλνουν, όπως σας έλεγα. Λοιπόν, Πόσο απρόβλεπτοι σε εισαγωγικά είμαστε εμείς ε, και ευνηδιαστικοί στους ε, ελέγχους μας. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Αν κυρίως βασιζόμαστε σε όσους ε, καταγγέλουν τα κακώς κείμενα και δεν βασιζόμαστε δική μας πρωτοβουλία, τότε είμαστε πολύ λίγο ευνηδιαστικοί, πολύ λίγο απρόβλεπτοι, οπότε κάποιοι κάνουν κάποιους άλλους να σιωπήσουν και να μην καταγγέλουν και τελειώνει η υπόθεση με τους ελέγχους. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω όσο σε ποιο ποσοστό των υποθέσεων δεν ξεκινούν μετά από κάποια καταγγελία. Ε, Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω στον κύριο Κέσλερ τη δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις και μετά θα γίνουν και ερωτήσεις στα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής. Οπότε θα δώσω τον λόγο στις δύο κυρίες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο κύριος Κέσλερ να μα μιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία και εγώ να σας συγχαρώ και να ευχηθώ καλή συνεργασία. Και τώρα θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εποπτείας για την εργασία που επιτέλεσε αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα θα ήθελα να μιλήσω για τον τρόπο που ε, ερμήνευσε η Επιτροπή Εποπτείας το ρόλο εγγύησης της ανεξαρτησίας της ε, Όλαφ. Νομίζω ότι το παράδειγμα που μας έδωσε αυτή η Επιτροπή μας βοηθά ιδιαίτερα. Όχι, όμως, όχι μόνο εμάς, αλλά και τη νέα Εποπτική Επιτροπή που αρχίζει το έργο της αυτές τις μέρες. Το... Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, παραγωγής, σκέψης και γνωμοδότησης της Επιτροπής αυτής ε, στα έξι χρόνια της λειτουργίας της. Δεν πρόκειται μόνο για ποσοτικό αλλά και για ποιοτικό έργο. Ξέρουμε τις ε, γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και νομίζω ότι αποτέλεσαν αυτά τα ε, δεδομένα τροφή για σκέψη όλων των ε, θεσμικών οργάνων. Καταρχήν, η Εποπτική Επιτροπή αναφέρθηκε σε μια συνεργασία που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή μεταξύ κρατών μελών. Η κατάσταση βελτιώνεται όπως είπε και η πρόεδρος Τεάτο, θα πρέπει να υπάρχει ένας κρατικός σύνδεσμος, ένας σύνδεσμος με τα κράτη για να έχουμε τάχιστα πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων και να μπορούμε να διενεργούμε και έρευνες τάχιστα. Και Δυστυχώς, κατά τις έρευνες είδαμε ότι δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ευτυχώς όμως έδωσε μία νέα όθηση συνεργασίας η Εποπτική Επιτροπή και χαιρόμαστε διότι το Κοινοβούλιο είναι πρωταγωνιστής αυτού του νέου κανονισμού 1073. Η Εποπτική Επιτροπή Επιτροπή μίλησε για την ανεξαρτησία της Όλαφ και θα πρέπει να δούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ερευνών όπως έγινε στο παρελθόν. Και πολλές φορές αμφισβητήθηκε η ανεξαρτησία ίδια της Όλαφ γιατί δεν μπόρεσε να διενεργήσει έρευνες όπως το επιθυμούσε και δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τους ισχύοντες κανόνες. Όχι μόνο τον ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Κοινοβουλίου. Έγινε λόγος και για την ατιμωρήσει, μάλλον έγινε λόγος για τις πολιτικές εντολές που έχουν οι ευρωβουλευτές. Και θα ήθελα να πω ότι μέσα στα πλαίσια αυτά υπάρχει και το θέμα ασυλίας των βουλευτών. γιατί πολλές φορές δεν μπορέσαμε ούτε να ε, μεταβούμε στα γραφεία μας. Για μερικούς ίσχυσε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ε, λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η εντολή μας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και δεν μπορεί να αναλυφθεί από την Όλαφ. Δεν μπορεί η Όλαφ να αλλάξει τους κανόνες, αλλά εφόσον εσείς είσαστε οι νομοθέτες, μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα δεδομένα. Επίσης, η Εποπτική Επιτροπή αποτάνθηκε στην Επιτροπή και έγινε λόγος για την πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων, στις τράπεζες δεδομένων της Κομισιόν και ε, ασχοληθήκαμε με το κατά πόσο θα πρέπει να ε, ανοίξουν έρευνες, να διενεργηθούν έρευνες ή να σταματήσουν δυσανάλογες έρευνες προσπαθούμε να φτάσουμε σε διευθετήσεις με την Κομισιόν, να δούμε ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί και πόσο μπορεί να μας βοηθήσει η Εποπτική Επιτροπή μέσα στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών για να υπάρξει και νομοθετική παρέμβαση εάν κριθεί αναγκαίο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Εποπτική Επιτροπή και να πω ότι η Επιτροπή αυτή εγγυάται την ανεξαρτησία της Όλαφ και βεβαίως προέβησε συστάσεις προς την ίδια την Όλαφ. Η Όλαφ μέσα στα πλαίσια μιας διάδρασης έλαβε υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα σε σχέση με τη διαδικαστική πορεία και την διαχείριση των ερευνών. Άρα, μετά από συστάσεις της Εποπτικής Επιτροπής, αλλάξαμε και ορισμένες διαδικαστικές διατάξεις. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι η Όλαφ αποστέλει τις τελικές εκθέσεις έρευνας σε όλα τα θεσμικά όργανα. Ιδιαίτερα όταν αμφισβητείται το κύρος ενός υπαλλήλου των θεσμικών οργάνων. Πρόκειται για το 1037, τον κανονισμό αυτό, άρθρο 9 του κανονισμού 1037. Εάν η έρευνα οδήγησε σε απόδοση ευθυνών, είτε οδήγησε σε απόδοση ευθυνών, είτε όχι και έτσι αποστέλλεται η τελική έκθεση στους εμπλεκόμενους ή στους ενδιαφερόμενους, ακόμα και αν ε, επί παραδείγματι ο βουλευτής κρίνεται αθώος μετά από διενέργεια μίας έρευνας. Είναι, πρόκειται για μια υποχρέωση, για διαφάνεια, για υποχρέωση διαφάνειας. Ε, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν δεν είχε δοθεί το σωστό follow-up. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εποπτική Επιτροπή και θα ήθελα να πω ότι οπωσδήποτε ε, δεν θα ε, αναγράφουμε τα ονόματα των πηγών μας. Θα διαγράφονται δηλαδή τα ονόματα των πηγών έτσι ώστε να μην τις εκθέτουμε. Επίσης κάτι άλλο που δεν εθίγει από την Επιτροπή αλλά από την εισηγήτρια θα ήθελα να πω ότι θα έχουμε θέματα συζήτησης αλλά δεν καταργήθηκε το τμήμα το οποίο ελέγχει τα στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία νομιμότητας, εσωτερική νομιμότητας. Δεν καταργήθηκε αυτό το τμήμα. Ε, καταργήθηκε το λεγόμενο Judicial Unit, το οποίο δεν ε, κρίνει την ε, νομιμότητα των πράξεων. Μιλάμε για την προστασία πηγών και δεδομένων. Τα, θέμα, τα θέματα της ασυλίας των ε, βουλευτών είναι θέμα το οποίο δεν αφορά τις δραστηριότητες της Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέσλερ για αυτά τα οποία μας είπατε. Πράγματι θα συνεχίσουν οι συζητήσεις ε, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Ευχαριστούμε για την ε, ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και πρέπει να γνωρίζουμε και να ζυγίζουμε τα διάφορα επιχειρήματα. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι η έκθεση της Εποπτικής Επιτροπής και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Και υπάρχει μια σειρά ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν να απαντήσουν νομίζω οι δύο ε, συντάκτε της έκθεσης. Γι' αυτό θα ήθελα να σα δώσω το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Για εμάς το τέλος της εντολής μας είναι πραγματικά α, ε, κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον το να ερχόμαστε εδώ πέρα και μπορούμε να αναφέρουμε τα πράγματα τα οποία παρατηρήσαμε και ε, το να έχουμε αυτή την επαφή με το Κοινοβούλιο χωρίς να επηρεάζουμε τον νομοθέτη απλά για να επισημάνουμε κάποια πράγματα τα οποία η Εποπτική Επιτροπή στη δραστηριότητα της ε, παρατήρησε και εκεί όπου υπάρχουν κάποιες ε, παρατηρήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές και να υιοθετηθούν. Γι' αυτό ευχαριστώ την κυρία Γκρέσλε για τα πολύ θεμελιωμένα ερωτήματά της, αλλά σας ευχαριστώ και για τους επένους τους οποίους επιδαψιλεύσατε στην Επιτροπή μας και οφείλω να πω πως ε, η εργασία αυτή στην Επιτροπή μας ε, χαροποίησε ιδιαίτερα. Τώρα για τα ερωτήματα, το θέμα του ελέγχου νομιμότητας, ε, ο οποίος αναφέρθηκε μαζί με μια επιθυμία που, έλε, που είχε πάντα η Επιτροπή μας, δηλαδή το προσωπικό των ελέγχων να ενισχυθεί. Στο παρελθόν ε, πάντα ένα 30% των εργαζομένων ασχολούνταν με τη βασική δουλειά του Όλαφ, αυτής έρευνες δηλαδή τώρα. Αυτό έχει αντιμετωπιστεί με το νέο οργανόγραμμα και έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ε, αυτός ο τομέας και ο κύριος Γενικός ε, Διευθυντής, ο κύριος Κέσλερ είναι αυτός ο οποίος το κατάφερε αυτό. Αυτό το βλέπετε και σε όλες τις γνωμοδοτήσεις μας για τον προϋπολογισμό που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και είναι σαφές πως λέμε πως πρέπει να ασχοληθεί με τη βασική του λειτουργία όλα. Βεβαίω, το θέμα μετά είναι τι γίνεται με αυτή την λεγόμενη ε, Judicial Unit και το πώς ε, εμπλέκεται σε έρευνες πώς θα λειτουργήσει αυτή η ε, συνεργασία. Δεν θα τολμήσω κάποια πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά οπωσδήποτε σημαντικό είναι να υπάρξει καλύτερη συνεργασία των διαφόρων μονάδων του Όλαφ. Τώρα, για όλα αυτά υπό τον όρο πως όπως είπα θα υπάρξει η σωστή συνεργασία τώρα. Όσον αφορά τους υπαλλήλους ε, κρατών μελών που ε, θα μπορούσε να προσλάβει ο Γενικός Διευθυντής, το ανέφερα και αυτό. Το ζήτημα λοιπόν ποιος κρίνει ε, αυτούς τους ανθρώπους ε, πρέπει να είναι κάποιος ο ανεξάρτητος δεν μπορεί να υπάρχει κάποια αυθαιρεσία ή να τους στέλνει απλά το κράτος μέλος χωρίς να ξέρουμε τι άνθρωποι είναι αυτοί αλλά το θέμα της νομιμότητας και των προσόντων είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί από κάποιον ανεξάρτητο και όχι ε, εντός ε, μιας ε, μονάδας. Το ζήτημα τώρα της ε, μετάδοσης των εκθέσεων χωρίς συνέχεια. Αυτό θα το αφήσω στην κυρία Ράιτ. Απλά θα ήθελα να πω πως οπωσδήποτε εδώ πέρα υπάρχουν παρεξηγήσει, αλλά υπάρχουν και σαφείς ε, διαφορές. Και όπως είπα στην αρχή, οι συστάσεις μας πρέπει να αποτελέσουν αφορμή έτσι ώστε ο νομοθέτης να σκύψει πάνω από αυτά τα ζητήματα και να δει υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα ή όχι. Και νομίζω αυτό ισχύει για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, για καταγγελίες ε, και έρευνες του Όλαφ εις ε, βάρος συγκεκριμένων θεσμικών οργάνων ε, και ευρωβουλευτών και την ασυλία που είναι πρωτογενές δίκαιο. Συμφωνώ πλήρως, αλλά πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, γιατί ο κανονισμός είναι ασαφής. Και ε, βεβαίως εδώ πέρα και εγώ φταίω γιατί είχα εμπλακεί στη σύνταξη του κανονισμού. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή και νομίζω και ε, για να απαντήσω τον κύριο Ρίμπιχ είναι ε, ένα θέμα προς διευκρίνηση αυτό στον κανονισμό. Νομίζω δεν έχουμε καμία διαφορά εδώ πέρα. Νομίζω λοιπόν κυρία Γκρέσλε πως απάντησα σε αυτά τα οποία είπατε και συμφωνώ πλήρως ε, με αυτά τα οποία αναφέρατε. Τώρα για τα υπόλοιπα θα συνεχίσει η κυρία Ράιτ. Για... Τον σκιοδησηγητή, ε, ναι, σας ευχαριστούμε. Τώρα, ε, κύριε Ρούμπιχ, ε, τα είπαμε για την ασυλία, για τις επαφές με τα κράτη-μέλη δεν είχαμε στο πλαίσιο της ε, εργασίας μας. Το ανέφερα παρενθετικά ως εμείς, ως Εποπτική Επιτροπή, δεν επιτρέπεται να παρέμβουμε στην διεξαγωγή των ερευνών. Η επαφή μας με τα κράτη-μέλη είναι έμεση, δηλαδή στο βαθμό που κάτι καταλήγει στις εθνικές δικαστικές αρχές. Κοιτάμε το εάν έχουν προστατευτεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία και αν εμείς ως εποπτική αρχή θα έπρεπε να κάνουμε μία επιπλέον έκθεση και δεν υπήρξε μία περίπτωση στην οποία θα έπρεπε να είχαμε κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα, το θέμα της διεύρυνσης αυτών των επαφών. Και αυτό είναι πάλι θέμα που ρυθμίζει ο κανονισμός. Εάν το θέλετε, εσείς ως νομοθέτης μπορείτε να δώσετε νέες τέτοιες δυνατότητες. Εγώ όμως θα ήθελα να πω μια που αναφέρθηκε η γραμματεία της Εποπτικής Επιτροπής. Εάν έχει νέες αρμοδιότητες η Εποπτική Επιτροπή, τότε θα πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό της. Ε, δεν μπορώ εγώ, και με συγχωρείτε για αυτή την προσωπική παρατήρηση, δεν μπορώ να φανταστώ πως τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής, τα οποία συνέρχονται ε, τουλάχιστον 10 ε, φορές ε, το χρόνο να παίρνουν ε, τις δουλειές τις, τους φακέλους σπίτι τους να το μελετήσουν. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται επίσης δεν είναι δυνατόν να κάνουν και αυτό το πράγμα παράλληλα. Ήταν δύσκολη δουλειά αλλά τα καταφέραμε. Νομίζω και το κάναμε πολύ ευχαρίστως. Τώρα για τη διαπίστωση για τους καταγγέλλοντες ε, θα τα απαντήσει αυτά η κυρία Ράιτ. Και για αυτούς είμαι μια καλύτερη ε, προστασία, αλλά αυτό θα ρυθμιστεί συνολικά ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει η Κομισιόν κάποιες προτάσεις. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην συνέχεια του έργου σας και είμαι σίγουρη ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Τεάτο. Πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Ράιτ, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και να πω πως δεν γράψετε μόνο ιστορία ως πρόεδρος της Επιτροπής μας, αλλά και στην Εποπτική Επιτροπή μαζί με τους ε, συναδέλφους σας. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Ράιτ. Thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ελάχιστα να προσθέσω σε αυτά που μας είπε η κυρία Τεάτο, αλλά ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις κυρίως από τον κύριο Σκυλακάκη σχετικά με το εύρος της απάτης και τι καλύπτεται από την αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία της Όλαφ. Όπως σωστά είπε ο κύριος Σκυλακάκης, δεν έχουμε καμία ιδέα, καμία εικόνα σε σχέση με την απάτη ως προς τον προϋπολογισμό. Ε, είναι μεγάλα τα μεγέθη, πελώρια, αυτό το ξέρουμε, ίσως... Κυρία Γκρέσλε θα μπορούσε Ε, συγγνώμη συνάδελφο να σας δώσει κάποιες ε, πληροφορίε σε σχέση με τον αριθμό των υποθέσεων. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στο ποσοστό των ερευνών που γίνονται βάσει καταγγελίας whistleblowing και πάλι εδώ δεν έχουμε εικόνα. Πάντως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Γκρέσλε και το Κοινοβούλιο σε σχέση με την υποστήριξή της ε, την υποστήριξη που όλο το Κοινοβούλιο μας προσέφερε για να υποστηρίξει το έργο της Εποπτικής Επιτροπής. Διευκολύνατε τα μάλλα το έργο μας ε, και Χαιρόμαστε πολύ που είχαμε τόσο καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύτιμη η βοήθειά σα. Το μπαλάκι τώρα είναι στο δικό σα γήπεδο και έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την κείμενη νομοθεσία του ώστε να διευκολύνετε την περαιτέρω το έργο τη Όλαφ και ο ρόλο μα ανέκαθεν δεν περιοριζόταν μόνο ε, στην κατοχήρεση τη ανεξαρτησία ε, των ελέγχων και τη Όλαφ αλλά και να υποστηρίζουμε το έργο τη Όλαφ, να τη διευκολύνουμε ώστε περισσότερε περιπτώσει ε, να καταλήγουν σε αίσιο τέλο. Λοιπόν, ελπίζουμε παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή τη ρότα. Ε, πάντως, ε, τη Δευτέρα όταν συναντηθήκαμε με τους ε, συναδέλφους της Νέας Επιτροπής, εντυπωσιαστήκαμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα σημειωθεί ραγδαία πρόοδος εφ' εξής και είμαστε όλοι τυχεροί που η Νέα Εποπτική Επιτροπή, η διάδοχός μας δηλαδή, θα είναι τόσο αποτελεσματική. Τα τελευταία έξι χρόνια εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά με την υποστήριξη και της δικής μας γραμματείας, με οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε σε σχέση με τη, αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλι ότι δεν είναι επαρκή η σύνθεση ε, της γραμματείας ούτως ώστε να έχουμε την απαιτούμενη γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, με τη νέα Εποπτική Επιτροπή αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο η έλλειψη επαρκούς τελέχωσης ε, δηλαδή καθώς και η, υποστή, η γραμματιακή υποστήριξη που υπάρχει. Προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα με τη βοήθεια της ε, κυρίας Γκρέσλα. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα κονδυλίων, διότι υπάρχουν, ε, ε, προβλέπονται κονδύλια ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την γραμματιακή υποστήριξη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πόσο ζωτικό είναι ο ρόλο ε, τη Εποπτική Επιτροπή και όπω σωστά είπε η κυρία Τεάτο, τα μέλη τη Επιτροπή ε, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δέκα φορέ συναντιούνται το χρόνο, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Είναι όλη η δουλειά που κρύβεται πίσω στην γραμματεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα μέλη τη Επιτροπή. Απευθύνω θερμότατη έκκληση ε, στο ε, βήμα της Επιτροπής σας, ούτως ώστε να ε, καταβληθούν σημαντικότερες προσπάθειες, ούτως ώστε να βελτιωθεί η στελέχωση της, της Εποπτικής Επιτροπής. Σχετικά με τις καταγγελίες, φυσικά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προωθήσουμε αυτές τις καταγγελίες. Υπάρχει και hotline στην Όλαφ, ούτως ώστε όσοι θέλουν να καταγγείλουν να αφήσουν μήνυμα. Δεν ήταν επανδρομένη αυτή η γραμμή αφήνανε μήνυμα λοιπόν οι καταγγέλλοντε και νομίζω ότι αυτό δεν έχει φέρει ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προτείνουμε λοιπόν να είναι επανδρομένη η υπηρεσία τηλεφωνική υποστήριξη για την ε, υποβολή καταγγελιών. Πιστεύω ότι θα αυτό θα ήταν πολύ αποτελεσματικό και θα υπήρχαν ε, πολύ περισσότερε πολύτιμέ πληροφορίε, ούτω ώστε η Όλεφ αυτεπαγγέλτο να ξεκινάει τι ερευνές τη. Δεν θέλω να σπαταλώ το χρόνο σα, Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάντω που μα ακούσατε. Σα ευχαριστώ για την ε, αυροφροσύνη σα και για την υποστήριξη που τόσο απλοχή μας προσφέρετε. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Ράιτ για την έκθεση και καθώς και για το έργο σας. Σίγουρα δεν σπαταλάτε εσείς το χρόνο μας, διότι μας απασχολεί πολύ το θέμα των ελεγκτικών μέτρων. Να γνωρίζουμε το η τώρα εντάσσεται στους ελέγχους για την καταπολέμηση της απάτης. Πέρα από τον έλεγχο όμως λειτουργεί ε, ως ελεγκτικός ε, φορέας σε άλλων οργάνων ε, ε, και πιστεύω ότι χρειάζεται και αυτό όπως ελέγχεται και η ίδια η Όλαφ, από άλλους. Οπότε θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας και θα ακούσουμε τώρα τις καταληκτικές παρατηρήσεις της κυρίας Γκρέσλε, αν έχει κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τις δύο κυρίες και το Γενικό Διευθυντή. Ένα πράγμα θέλουμε να εμποδίσουμε, να μην γίνει όλα ξανά ο αυτό το οποίο είχαμε. Έχουμε όλοι κακές αναμνήσεις. Δεν θέμε ξανά κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικός ο διοργανικός χαρακτήρας του Όλαφ και είναι σημαντικό οι εσωτερικές έρευνες να μην ε, εμποδίζονται από διάφορα μέτρα. Αυτό είπαμε και γι' αυτό βεβαίως είναι πολύ σημαντικές οι συστάσεις της Εποπτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και δώστε τους χαιρετισμού μας και στα υπόλοιπα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, τελειώσαμε και με αυτό το σημείο της ε, μέρης διάταξης. Ευχαριστούμε την κυρία Τεάτο, την κυρία Ράιτ και τον Γενικό Διευθυντή του Όλαφ και περνάμε άρα στα διάφορα. Δεν υπάρχουν τίποτα. Εκεί πέρα. Επόμενη συνεδρίαση 9 Φεβρουαρίου την Πέμπτη και έτσι τελειώνει το δημόσιο μέρος της συνεδρίασης. Να υπενθυμίσω στους συντονιστές πώς έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων.